Well, thank you very much. Good morning and uh, let... Καλημέρα. Να συνεχίσουμε τις συζητήσεις μας για την κατάσταση στο Μαλί και θα ήθελα ε, το μικρόφωνο Θα ήθελα λοιπόν να παρουσιάσω τον κύριο Νίκολας Βέστχολτ, που είναι ο ασκόν ε, ε χρέη διευθυντού στην υπηρεσία εξωτερικής δράσης και ο κύριος Στίβενς που είναι επίσης στην ίδια υπηρεσία, ο υπονάβαρχος Μπρουσ Βίλιαμς που είναι αναπληρωτής επικεφαλής του στρατιωτικού επιτελείου. Δίνω το λόγο στον κύριο Ντανζόν. Ευχαριστώ Ιωάνν, καλημέρα. Ευχαριστώ που είστε εδώ μαζί μας σήμερα το πρωί για το καυτό θέμα της στιγμής. Δεν θα επανέλθω σε όσα υπόθηκαν για το πόσο σοβαρή και πήγουσα είναι η κατάσταση στο Μαλί. Όλοι έχουμε συνέστηση. Το έχουμε συζητήσει επανειλημμένα, εκπλησόμενοι από τότε, παρά τις προειδοποίησεις παρά τις απειλές που είχαν σαφώς ανιχνευθεί παρά την ομοφωνία που υπάρχει στην Ένωση για το θέμα αυτό και που μας είχαν ε, οδηγήσει στο να υιοθετήσουμε μια στρατηγική για το Σαχέλ σήμερα δίνουμε την εντύπωση ότι εξεπλάγημεν όλοι οι Ευρωπαίοι δυσάρεστα εξεπλάγημεν χθες με τον Πατρίκ Ντερουζιέ, τον πρόεδρο της ε, Στρατιωτικής Επιτροπής και μετά με τον αντιστράτηγο Ρουμπί που ήταν εκπρόσωπος ε, της Ένωσης, στρατιωτικός της Ένωσης. Συζητήσαμε τα τρέχοντα θέματα. Τώρα θέλουμε να δούμε σφαιρικά το θέμα αυτό. Θα γίνει, ή μάλλον έγινε, στις 17 Ιανουαρίου ένα έκτακτο Συμβούλιο Υπουργών Εξωτερικών και υιοθέτησε οκτώ πορίσματα εκ των οποίων το πιο ουσιώδες και ορατό είναι το e UTM Mali, αυτή η αποστολή εκπαίδευσης που εδώ και κάποιους μήνες ε, σκοπεύαμε να την ε, υλοποιήσουμε. Υπάρχουν και χρηματοδοτικές πλευρές, η χρηματοδότηση της αφρικανικής δύναμης που θα αναπτυχθεί και επίσης η πολιτική διαδικασία, γιατί έχουμε συνέστηση ότι ναι μεν προτεραιότητα τώρα δίδεται στις στρατιωτικές επιχειρήσεις αλλά ότι όλα αυτά εάν δεν συνοδευτούν σύντομα από μια πολιτική διαδικασία δεν θα οδηγήσουν σε ουσιώδη αποτελέσματα. Η Ένωση έχει αρκετά μέσα, ε, αρκετές δυνατότητες, αρκετούς μοχλούς όμως ε, λυπούμεθα που δεν αξιοποιήθηκαν όλες αυτές τις δυνατότητες για να προλάβουμε την κρίση. Δεν αξιοποιήθηκαν νωρίτερα. Είμαι αρκετά επικριτικό επ' αυτού, του θέματος, αλλά στόχος είναι τώρα να δούμε το μέλλον, όχι να αποτιμήσουμε το παρελθόν, τα γεγονότα. Ο επίγον χαρακτήρας είναι σαφή. Πρέπει να ανακτήσουμε την πρωτοβουλία, γιατί η κατάσταση όπως είναι τώρα αν δεν θεωρηθεί αποτυχία, θα πρέπει να θεωρηθεί καθυστέρηση αντιμετώπισης. Αυτά λοιπόν είναι τα κύρια στοιχεία. Να δώσω πρώτα απ' όλα το λόγο στον Νίκολας Βέστκοτ, Γενικό Διευθυντή για την Αφρική. Ευχαριστώ. Θα προτιμήσω να αφήσω πολύ χρόνο στις ερωτήσεις σας. Βεβαίως ε, είμαι σίγουρος ότι ξέρετε την ε, κατάσταση επιτόπου και για ποιο λόγο επεμβαίνει η Ένωση. Υπήρξαν δραματικές εξελίξεις από την αρχή του μήνα και χρειάστηκε να αντιδράσουμε ως δυνατόν συντομότερα. Οι δυνατότητες ε, των Γάλλων ε, επέτρεψαν να αντιδράσουν ε, στιγμιαία, αμέσως, για να σταματήσουν τις δυνάμεις των ανταρτών που προχωρούσαν προς τον Μπαμάκο. Και η Ένωση εξέφρασε και την ε, άποψή της κατά το έκτακτο Συμβούλιο Υπουργών Εξωτερικών που συνεκάλεσε η κυρία Άστον 17 Ιανουαρίου. Τώρα, θέλω να σε ενημερώσω για το πώς εφαρμόζουμε τα πορίσματα αυτού του έκτακτου, έκτακτου Συμβουλίου Υπουργών Εξωτερικών και ποια είναι τα επόμενα βήματα πέρα από τα συμπεράσματα για να επιχειρήσουμε να επιλύσουμε την κρίση στο Μαλή, ειδικά στο Σαχέλ γενικότερα. Γιατί η περιφερειακή διάσταση πρέπει να είναι σαφή καθ' όλη τη διάρκεια τη αντιμετώπιση μαζί Η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης, αναλαμβάνοντα αυτέ τι ενέργειε ενέργειες, στοχεύει στην προστασία των στρατηγικών συμφερόντων και συμφερόντων ασφαλείας της Ένωσης, αυτή καθεαυτή, που απειλούνται από την αποσταθεροποίηση του Σαχέλ και δεύτερον να υποστηρίξει το λαό του Μαλή επιτρέποντας σε όλους τους ε, πολίτες του Μαλή, σε όλη την επικράτεια του Μαλή, να έχουν τη δυνατότητα να επιλέξουν την ε, κυβέρνηση της επιλογής τους και να ζουν εν ειρήνη και ευημερία ε, με τους λογικούς πόθους τους για ανάπτυξη και ειρήνη. Πόθους τους για ανάπτυξη και ειρήνη που κατοχυρώνονται στο σύνταγμά τους και όλα αυτά τα ιδεώδη ένα μεγάλο τμήμα του λαού του Μαλή αυτή τη στιγμή δεν είναι σε θέση να τα απολαύσει. Αυτές είναι οι αρχές που είναι βάθρο της επέμβασής μας. Όπως ξέρετε εφαρμόζουμε και τα διδάγματα από προηγούμενες κρίσεις στην Αφρική προσπαθώντας να έχουμε μια ολοκληρωμένη προσέγγιση. Το θέμα της ασφάλειας είναι βέβαια το πιο σημαντικό, η στρατιωτική δράση που έχει αναλυφθεί για να αποκαταστήσει τον έλεγχο στην επικράτεια του Μαλή. Εγώ θα πω λίγα λόγια γι' αυτό. Ο Walter Stevens και άλλοι συνάδελφοι θα πούν περισσότερα. Δεύτερον, ωστόσο και εξίσου σημαντικό, υπάρχει μια πολιτική, όπως είπα, διάσταση στην προσπάθεια εξέβρεσης λύσης. Να δημιουργήσουμε δηλαδή, να οικοδομήσουμε μια πιο στεναρή δημοκρατία για το λαό του Μαλή, να τους βοηθήσουμε να έχουν μια πιο σταθερή δημοκρατία που να μπορεί να υπερασπιστεί τον εαυτό της και όπου όλες οι ομάδες της χώρας να έχουν το αίσθημα ότι η φωνή τους γίνεται ακουστή και ότι μπορούν να συμμετάσχουν. Δεν είναι κεραυνός ενεθρία η κρίση στο Μαλί. Υπήρξαν δυσχέρειες παντού στο Σαχέλ. Η ένταξη κάποιων ομάδων, του και άλλες ομάδες και άλλες μειονότητες δεν ήταν πάντα ευχερής. Υπήρξαν διαδοχικές ανταρσίες, ε, συγράξεις και εμφύλοι πόλεμοι από την ανεξαρτησία. Αυτή ωστόσο είναι η πιο σοβαρή και η πιο δραματική λόγω των επιδράσεων και στον υπόλοιπο κόσμο. Μας δίνει ωστόσο την ευκαιρία να επιχειρήσουμε να οικοδομήσουμε πολιτικές δομές που να είναι πιο ανθεκτικές για να οικοδομηθεί στο Σαχέλ πιο μακροπρόθεσμη σταθερότητα. Αλλά αυτό μπορεί να συμβεί μόνο εάν υπάρχουν και κάποιες ε, λογικές προοπτικές ανάπτυξης. Βεβαίως παρέχουμε ανθρωπιστική βοήθεια για να επιβιώσουν οι πληθυσμοί, ιδιαίτερα όταν μετατοπίζονται από τις αιστείες τους, αλλά ελπίζουμε να έχουμε τη δυνατότητα και μακροπρόθεσμα να ενισχύσουμε την ανάπτυξη της περιοχής, ούτως ώστε να υπάρχουν ευκαιρίες και για τους νέους. Πρώτον, για την ασφάλεια. Θα επιταχύνουμε τις προσπαθειές μας ούτως ώστε να υποστηρίξουμε τις γαλλικές και μαλλικές δυνάμεις. Μέσω αυτής της αποστολής των Ηνωμένων, ε, μέσω αυτής της για την εκπαίδευση και επίσης μέσω ε, της άλλης ε, της αφρικανικής δύναμης που θα αναπτυχθεί στο Μαλί η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει δεσμευτεί να χορηγήσει για αυτήν την αφρικανική προσπάθεια οικονομική βοήθεια, χρηματοδότηση. Ο Επίτροπος Πίμπαλξ είπε ότι έχουμε διαθέσιμα 50 εκατομμύρια ευρώ για αυτή την προσπάθεια και θα συμμετάσχουμε και στην ε, συνδιάσκεψη των δωρητών που θα γίνει στα πλαίσια τη Αφρικανική Διάσκεψη Κορυφή στην Αντίσα Μπέμπα 29 Ιανουαρίου. Θα συμμετάσχουμε με διάφορου άλλου εκπροσώπου τη Ένωση για να συζητήσουμε πώ θα συμβάλλουμε και θα συνδυάσουμε την ε, βοήθειά μας με άλλα μέλη της διεθνούς κοινότητα, τα Ηνωμένα ΕΕ, Έθνη, Ηνωμένε ΗΠΑ και άλλου ενδιαφερόμενους. Οι προσπάθειε της Αφρικανικής Ένωσης και των κρατών μελών τη και των χωρών που είναι στο ΕΚΟΟΑΣ και των χωρών που είναι εκτός της ΕΚΟΟΑΣ επίσης θα συμβάλλουν σε αυτή την προσπάθεια για να επανέλθει η ασφάλεια και η σταθερότητα στο Μαλί. Βεβαίω μπορούν και τα κράτη-μέλη της Ένωσης, να συνάδελφοι θα σα πούν τι άλλες ιδέες υπάρχουν, για παράδειγμα, να υπάρξει μια κεντρική μονάδα ανταλλαγής ε, παρεμβάσεων και συμβολών. Στην ε, συνεδρίαση των Υπουργών Εξωτερικών στι 17 Ιανουαρίου μας ενημέρωσε ο Υπουργό Εξωτερικών του Μαλή, ο κ. Κουντιβάλη. Μα ε, του καταστήσαμε σαφέ ότι η υποστήριξη τη Ένωση βασίζεται στην προσπάθεια να υπάρξει δημοκρατική και συνταγματική αποκατάσταση στο Μαλί. Και γι' αυτό λοιπόν ο δικός χάρτης προς αυτήν την κατεύθυνση είναι ουσιώδες ε, στοιχείο για να θεωρήσουμε ότι είναι λογικό να υποστηρίξουμε τις δυνάμεις του Μαλή μέσω αυτής της αποστολής εκπαίδευσης και γενικότερα στην προσπάθεια να αποκατασταθεί η ενότητα της χώρας. Καταλαβαίνουμε ότι ο δικός χάρτης ε, είναι ακόμη υποσυζήτηση, θα πρέπει να εγκριθεί από το Συμβούλιο των Υπουργών της προσωρινής κυβέρνησης υπό τον Πρόεδρο Ταωρέ και θα υποβληθεί στην Εθνική Συνέλευση, στην Εθνοσυνέλευση και ελπίζουμε μέσα στο επόμενο 10 πενθήμερο να υποβληθεί. Δεν θα είναι, μια, δεν θα είναι ένα συνολικός δικός χάρτης, δεν θα περιέχει όλα όσα θα θέλαμε, αλλά στόχος είναι να εκινήσει η διαδικασία μια διαδικασία που θα επιτρέψει να συμμετάσχουν όλες οι πολιτικές δυνάμεις στη χώρα, ούτω ώστε να αποκατασταθεί κάποιο είδος δημοκρατικής κυβέρνησης που να είναι υπόλογη στον πληθυσμό της χώρας. Επίσης, θα γίνει μια συνεδρίαση της ε, ομάδας για την παρακολούθηση της κατάστασης στο Μαλή εδώ στις Βρυξέλλες στις 5 Φεβρουαρίου. Θα τη φιλοξενήσουμε εμείς ως Ένωση. <clears throat> θα αξιοποιήσουμε αυτή την ευκαιρία για να συζητήσουμε με τους εκπροσώπους της κυβέρνησης του Μαλή πώς θα στήριξουμε την εφαρμογή αυτού του οδικού χάρτη που είναι πολύ σημαντικός για το μέλλον της χώρας. Πρέπει να είναι στεναρή αυτή η διαδικασία για να μπορέσουμε να τους υποστηρίξουμε κατά την εφαρμογή του οδικού χάρτη. Τώρα, η πλευρά της ανάπτυξης. Το Μαλί, όπως ξέρετε, πέρασε μια πολύ τραυματική εμπειρία, έχει περιορισμένα μέσα. Τα θεσμικά όργανα του κράτους, οι θεσμοί, έχουν αρχίσει να καταραίουν. Παράλληλα λοιπόν με τον οδικό χάρτη πρέπει να επιτρέψουμε να, λειτουργού, να, επιτρέψουμε να συνεχίσουν να λειτουργούν οι θεσμοί του κράτους. Τα σχολεία πρέπει να είναι ανοιχτά και να διδάσκουν. Θα πρέπει να υπάρχουν υγειονομικές υπηρεσίες που να παρέχουν υγειονομικές υπηρεσίες στους κατοίκους της χώρας. Πρέπει να συνεχιστούν κάποια προγράμματα ώστε να υπάρξει μια κάποια επιστηστική ασφάλεια, μια κάποια ανθεκτικότητα. Θα στείλουμε λοιπόν μια αποστολή από διάφορες υπηρεσίες της Ένωσης στον Μπαμακό προσεχώς για να αποτιμήσουμε τις ανάγκες τους, να συζητήσουμε με την κυβέρνηση, να δούμε τι χρειάζεται. Η περισσότερη από την αναπτυξιακή μας βοήθεια προς την κυβέρνηση έχει ανασταλεί από το πραξικόπημα. Τώρα θέλουμε να εξετάσουμε αν μπορεί να ξαναρχίσει ένα τμήμα της, αλλά πρέπει να είναι πολύ καλά στόχο προσιλωμένη και να εντάσσεται στα πλαίσια της πολιτικής διαδικασίας που περιέγραψα. Πρώτο βήμα λοιπόν είναι να δούμε τι ακριβώς χρειάζονται, πού χρειάζονται τη βοήθειά μας να τους στηρίξουμε με τον πιο επωφελή τρόπο αυτήν την ε, προσωρινή κυβέρνηση με τον ε, Πρωθυπουργό Σισόκο. Με αυτούς θέλουμε να συζητήσουμε. Αυτές είναι οι τρεις ε, ενέργειες που προβλέπουμε για το εγγύς μέλλον. Η Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης προσπαθεί να συντονίσει τις ενέργειές της με την Επιτροπή, με τους στρατιωτικούς μας, με όλες τις γενικές διευθύνσεις της Επιτροπής που ε, εμπλέκονται. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ κύριε Πρέσβη. Ο κύριος Στίβενς. Έξι σημεία. Σε ό,τι αφορά την ε, αποστολή ε, κατάρτισης του Μαλικού στρατού. Καταρχάς, το πρώτο σημείο είναι σύντομο. Η αποστολή UTM έχει σαν σκοπό να καταρτήσει τον στρατό. Είναι τμήμα μιας ευρύτερης προέγγισης, το πολιτικό τμήμα, το ανθρωπιστικό τμήμα, το ανταπτυξιακό τμήμα, αλλά και το τμήμα της ασφάλειας είναι τμήματα αυτής της προσπάθειας. Δεύτερον, ε, σχεδιάζουμε εδώ και αρκετό καιρό αυτή την αποστολή και μετά τις τελευταίες ε, εξελίξεις ε, άλλαξαν τα δεδομένα. Αλλά δεν άλλαξε η ουσία της αποστολής. Παραμένει ο στόχος αποστολής ο ίδιο. το μαλλί χρειάζεται κατάρτιση, χρειάζεται αναδιάρθρωση, ε, τώρα περισσότερο παραποτέ. Φυσικά θα πρέπει να δούμε κάποιε κάποιες λεπτομέρειες, δηλαδή πώς θα διαρθώσουμε την εκπαίδευση. Ή, θέλαμε να εκπαιδεύσουμε τέσσερις ομάδες μάχης ε, σε όλες τις τεχνικές, να δούμε όμως και την διοικητική αλυσίδα, να διαρθώσουμε το στρατό. Θα θέλαμε να δούμε και κάποιες μονάδες στρατού οι οποίες θα πολεμήσουν στο μέτωπο. κάποιες από αυτές τις, ε, κάποια από αυτά τα θα πρέπει να δώσουν μάχες, θα πρέπει να μπορούν να δώσουν μάχες. Θα πρέπει να δούμε και την τοποθεσία ε, της ε, αποστολής που θα λάβει η χώρα στο Σέγκο, 250 χιλιόμετρα βόρειο ανατολικά από τον Παμάκο. θα χρησιμοποιηθεί επίσης και από τις γαλλικές δυνάμεις αυτή η αποστολή ή μάλλον αυτή η αποστολή έχει χρησιμοποιηθεί, αυτό, η τοποθεσία η ε, χρησιμοποιηθεί από το γαλλικό στρατό και τώρα θα πρέπει να βρούμε μια άλλη τοποθεσία. Όλα αυτά τα στοιχεία θα πρέπει να τα ενσωματώσουμε στο σχεδιασμό της αποστολής. Ετοιμάζονται οι διοικητές. Ο στόχος παραμένει ο ίδιος, να εκπαιδεύσουμε και να αναδιαφρώσουμε το στρατό του Μαλή και να τον καταστήσουμε αποτελεσματικό υπό τον έλεγχο των πολιτικών δυνάμεων και των δημοκρατικών δυνάμεων της χώρας. Έχουμε επιταχύνει τις διαδικασίες και αυτό σημαίνει ότι το Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων την ε, περασμένη Πέμπτη ε, αποφάσισε για την αποστολή, διόρισε τον ε, διοικητή, τον στρατηγό Le και στείλαμε μία ομάδα ήδη υπεύθυνους για την επιμελητία, για την υποδομή, μια μικρή ομάδα, καθώς και άτομα τα οποία ε, θα προετοιμάσουν την αποστολή. Η Πολιτική Επιτροπή και η Πολιτική ε, Επιτροπή Ασφαλείας είναι υπεύθυνοι. Οι υπεύθυνοι θα έρθουν ε, στην Επιτροπή αυτή και θα λογοδοτήσουν. Θέλουμε να ξεκινήσουμε την αποστολή στις 12 Φεβρουαρίου και η ανάπτυξη των... της αποστολής αυτής θα ακολουθήσει τις επόμενες μέρες. Αυτό μου λέει ο διοικητής της ε, αποστολής. Μου λέει ότι δηλαδή αμέσως μετά μπορούμε να αρχίσουμε την εκπαίδευση. Το πέμπτο σημείο είναι σημαντικό. Συνδέεται με τον εξοπλισμό του στρατού του Μαλή. Εμείς θα καταρτήσουμε το στρατό του Υπάρχει το θέμα της επιμελητίας, του εξοπλισμού, του στρατού και θα καταβληθούν πολλές προσπάθειες, θα χρειαστούν πολλές προσπάθειες πέρα από αυτά που κάνουμε για να υποστηρίξουμε την αφίσμα. Θα ήθελα να σας επιστήσω την ε, προσοχή ότι στις 29 Ιανουαρίου θα γίνει στην ε, Αντίς Αμπέμπα ε, μία διάσκεψη των δωρητών και θα συζητήσουμε και αυτό το θέμα. Υπάρχει δυνατότητα εκεί η UTM να συντονίσει την αποστολή. Θα κοιτάξουμε και τις ε, διμερείς επαφές με άλλους δωρητές. Ε, θα πρέπει βεβαίως να κινητοποιηθεί η διεθνής κοινότητα γι' αυτό. Και όπως είπε και ο Νίκ, ε, υπάρχει η Επιτροπή Παρακολούθησης που θα συνεδριάσει στις 5 Φεβρουαρίου εδώ για το θέμα αυτό. Είναι σημαντικό αυτό το θέμα, πέρα από την υποστήριξη προς την αφήσμα ο ναύαρχος ε, Williams θα σας πει και κάποια πράγματα για το γραφείο συμψηφισμού. Μας απασχόλησαν τα προβλήματα στην, ε, στο Σαχέλ, στο Νίγηρα, στο, στις υπόλοιπες χώρες. Υπάρχει μια αποστολή που βοηθάει τις ε, δυνάμεις του Νίγηρα για να καταπολεμήσουν τις εγκληματικές ομάδες οι οποίες συνδέονται με τρομοκρατικές δραστηριότητες και λέγεται UCAP Niger. Είναι μια πολιτική αποστολή με στρατιωτικά στοιχεία και βοηθάει τις δυνάμεις του Νίγηρα να καταπολεμήσουν την τρομοκρατία και τις εγκληματικές ομάδες. Έχει και περιφερειακά στοιχεία. Έχει ένα αξιωματικό συνδέσμου στον Παμάκο και θα ενισχύσουμε ε, την σύνδεση αυτή στον Παμάκο, ούτως ώστε να βοηθήσουμε και τις δυνάμεις του Μαλή να καταπολεμήσουν την τρομοκρατία και τις εγκληματικές ομάδες. Και θα επεκτείνουμε την αποστολή στον Νίγηρα. Ε, μάλιστα, είχαμε προτείνει την ίδια αποστολή στις αρχές του Μαλή που δεν συμφώνησαν. Θα την επεκτείνουμε και στο Μαλή, λοιπόν, ούτως ώστε να καλύψουμε τη Σαχέλ, θα καλύψουμε μάλιστα και τη Μαυριτανία. Για τις α, ομάδες μάχης, α, μπορώ να σας πω κάποια στοιχεία, αν μου θέσετε ερωτήσεις. Ευχαριστώ. Κύριε Πρέσβη, Ναύαρχε Μπρούς Βίλιαμς, είστε ο αναπληρωτής διευθυντής της Γενικής Δύναμης Ευρωπαϊκής Ένωση, σα ευχαριστούμε που είστε εδώ. Μάλιστα σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα απαντήσατε στην πρόσκλησή μας και έχετε το λόγο. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Δύο λόγια θα ήθελα να σας πω για να προσθέσω στα όσα είπαν οι συνάδελφοι. Το θέμα της εξέβρεσης αφρικανικής λύσης σε ένα αφρικανικό πρόβλημα σημαίνει ότι το στοιχείο στήριξης που υποδείχθηκε θα πρέπει να περιλαμβάνει όλα τα στοιχεία της ε, διοικητικής μέρημνας που θα μπορέσει να βοηθήσει την αφίσμα, τις αφρικανικές δυνάμεις δηλαδή, να ανταποκριθούν σε αυτή την εντολή. Ο στόχος της δημιουργίας ενός καθαριστικού κέντρου, θα λέγαμε, στην ουσία θεωρήθηκε πως θα λειτουργήσει ως καταλήτης για την στήριξη αυτή τη διοικητικού τύπου που ανέφερε το Συμβούλιο την περασμένη εβδομάδα. Το πρόβλημα με κάθε αναδυόμενη κρίση είναι να μπορέσουμε να συγκεντρώσουμε τις απαιτήσει με δυνητικούς δωρητές, αλλά και αντιστρόφως ανάλογα να κατανοήσουμε τι θα επιθυμούσαν να δώσουν οι δωρητές και μετά αυτά να τα αντιστοιχίσουμε με τις ε, ανάγκες. Ο στόχος αυτού του καθαριστικού κέντρου, θα έλεγα, είναι να λειτουργήσει ως καταλήτης, δηλαδή να διευκολύνει, να συντονίσει, να συγκεντρώσει, να ελέγξει και να ιεραρχήσει τις απαιτήσει της αφίσμα, ώστε να την βοηθήσει να μπορέσει να έχει τον κατάλληλο εξοπλισμό που χρειάζεται για να ανταποκριθεί στο έργο που έχει να κάνει στο Μαλί. Αμέσως μετά από το Συμβούλιο της περασμένης εβδομάδας ξεκινήσαμε και αυτό βασίζεται σε ένα αρκετά απλό σύστημα, όπου δηλαδή το κέντρο του συντονιστικό ε, βρίσκεται στο στερεωτικό προσωπικό της Ευρωπαϊκής Ένωσης και βασίζεται σε αξιωματικού σύνδεσης στις χώρες ε, που ένας βρίσκεται στα επιτελείο της ECOWAS και Στόχο έχει να βοηθήσει και να αποτελέσει μέλος των παφών και των προβληματισμών της αφίσμα από, την, από το περασμένο έτος και ο άλλο μέλος, ο άλλος οκτηματικός σύνδεσης θα είναι στην Μπάμακο, ε, στο επιτελείο της αφίσμα εκεί. Στόχος είναι λοιπόν να ενθαρρύνουμε τα κρατημέλη να χρησιμοποιήσουν αυτές τις δυνατότητες για να συντονίσουν τη συμμετοχή τους, την ανταπόκρισή τους και από εμά να μπορέσουμε να συγκεντρώσουμε από την ΕΚΟΒΑΣ, από την αφίσμα και από τους υπόλοιπους τις ανάγκες τους όσον αφορά την ε, στήριξη την διοικητική και την ηλική. Στην ουσία πρόκειται για ένα είδος προξενιού, όπου βάζουμε δηλαδή από τη μια πλευρά τον δωρητή και από την άλλη πλευρά τον αποδέκτη της δωρεάς. Έχουμε την αφίσμα και, το, και ένα κράτος μέλος της αφίσμα που θα συλλέξει την δωρεά, ώστε να έχουμε δηλαδή όσο γίνεται πιο γρήγορη στήριξη. Αυτός είναι ο στόχος του καθαριστικού αυτού ε, ε, οίκου, κέντρου θα λέγαμε, ένας, ε, μια διευκόλυνση μια διαδικασία όμως που έχει ξεκινήσει από τις αρχές του περασμένου έτους για να προσπαθήσουμε να διευκολύνουμε τις διαδικασίες της ECOWAS για να αναπτύξει την αφίσμα της Αφρικανικές Στρατιωτικές Δυνάμεις για να φέρει σε πέρα στο έργο που έχει αναλάβει στο Μαλί. Ευχαριστούμε. Ναύαρχε, πριν να δώσω το λόγο στους συναδέλφους, θα ήθελα εγώ να επανέλθω σε κάποια σημεία. Κατά τη διάρκεια της έκτακτης σύσκεψης του Συμβουλίου των Υπουργών Εξωτερικών της 17ης Ιανουαρίου, από τα οκτώ σημεία των συμπερασμάτων, είχαμε την ευκαιρία να το πούμε, τελικά τα επτά ήταν σημεία που ήδη είχαν κατά κάποιο τρόπο προετοιμαστεί ή συμφωνηθεί κιόλα, δηλαδή το Συμβούλιο παρακολούθησε μια επιτάχυνση μάλλον, μάλλον ε, βοήθησε στην επιτάχυνση απέναντι στην ε, επίγουσα κατάσταση, ωστόσο αναφέρθηκε ο διορισμός ενός ειδικού εκπροσώπου για το Σαχέλ. Πέρα από το γεγονό ότι δεν είμαι πεπισμένο πω αυτό θα είναι η κατάλληλη απάντηση, αλλά εν πάση περιπτώσει αυτό είναι άλλο θέμα. Το... Πού βρισκόμαστε με αυτή τη διαδικασία, Ήδη κυκλοφορούν κάποια ονόματα. Είναι κάποιος ήδη έτοιμος να φύγει. Θα ήταν μάλιστα ενδιαφέρον να δούμε πώς αυτός ο άνθρωπος θα συνεργαστεί με τον κύριο Πρόντι που είναι ο ειδικό εκπρόσωπος ε, των Ηνωμένων Εθνών και που γνωρίζει πολύ καλά τα ευρωπαϊκά γρανάζια. Θα έχουμε δύο ανθρώπους ε, λοιπόν και θα είναι ενδιαφέρον να δούμε ποιοι θα είναι αυτοί και ποιο είναι το προφίλ τους. Και έπειτα η ερώτηση που μου έρχεται τελείως αυτόματα είναι το θέμα των ε, μάχημων μονάδων. Ξανά και ξανά, over and over όπως λέμε στα γαλλικά. Το έχουμε πει και ξαναματαπεί. Σε τι χρησιμεύει αυτή η υπέροχη εφεύρεση που στην ουσία για την ώρα είναι απλώς εικονική. Έχουμε δηλαδή φέτος ε, ένα battle group, μια με μονάδα κρούσης που αποτελείται από στρατιωτικούς της Γερμανίας, της Γαλλίας, της Ολλανδίας λοιπά μέσα στο πλαίσιο της κοινή ευρωπαϊκής πολιτικής άμυνας και ασφάλειας, μιας πολιτικής που θέλουμε να αναπτύξουμε απέναντι σε μια κρίση που καλεί που ε, καλεί σε δράση την ε, ομάδα κρούσης που αποτελείται από Γερμανούς, είπα, Μεγάλους και Πολωνούς και η οποία είναι ανύπαρκτη. Υπάρχει, δεν υπάρχει. Αν υπάρχει, γιατί δεν παρεμβαίνει. Ε, πώς μπορούμε να εξηγήσουμε ότι στην ουσία έχουμε ένα και σπάνιο συλλογικό μέσο στη διάθεσή μας, το οποίο όμως δεν λειτουργεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτά και δίνω το λόγο αμέσως στον Μάικλ Γκάλερ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ευχαριστώ για τα εισαγωγικά που ακούσαμε. η στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το Σαχέλ που δεν είναι τόσο πρόσφατη υπάρχουν μια σειρά από δυνατότητες ορισμένες ήδη αναφέρθηκαν καμιά φορά εκπλήσωμε από την έκπληξη που προκάλεσαν κάποιες εξελίξεις ήδη από την κατάρρευση του καθεστώτος ε, Καντάφη ξέραμε ότι κάποιες δυνάμεις από τη Λιβύα δεν ήταν μόνο πια στα βόρεια του Μαλία, αλλά σιγά σιγά σε ολόκληρη την περιοχή και είχαν αναλάβει τον έλεγχο ορισμένων περιοχών. Όπως είπα και χθε, διερωτώ με, γιατί ξέρετε ότι στις 15 Οκτωβρίου ήδη αποφασίστηκε αυτή η αποστολή εκπαίδευσης της ε, Ένωσης και αν θυμάμαι είχαμε μιλήσει για επιτάχυνση των διαδικασιών διερωτώ με τι έγινε αυτούς τους τρεις μήνες ή μάλλον τι δεν έγινε. Γιατί ακόμη δεν έχουμε προχωρήσει αρκετά. Γιατί θα μπορούσε να γεννηθεί η υποψία ότι κάπου κάποιος μυστικά ε, θεωρούσε ότι μπορεί να το θέμα αυτό να ρυθμιστεί από μόνο του, ότι μπορούν κάπως όλοι αυτοί οι τζιχάντες να σταματήσουν να προελάβουν. Όμως συνέχισαν. Δεν με ικανοποιεί λοιπόν ε, ο ρυθμό με τον οποίο εφαρμόστηκαν ε, αυτά που αποφασίσαμε γιατί δεν είναι δυνατόν να θεωρεί κανεί ότι εξεπλάγει από τι εξελίξει. Συγκεκριμένα τώρα, οι διάφορες μονάδες, τα διάφορα εξτρατευτικά σώματα. Ναι βεβαίω θα υπάρξουν αφρικανικές δυνάμεις που ποτέ δεν έχουν συνεργαστεί μέχρι στιγμής. Ποτέ δεν έχουν αναπτυχθεί μαζί. Θα είναι σε θέση ταυτόχρονα να εκπαιδευτούν, να ε, μπορέσουν να συνεννοηθούν. Γιατί θα πρέπει ε, να υποστηρίξουν ε, σε μάχες τον στρατό του Μαλή. Για τον οποίον στρατό του Μαλή έχουμε υπόψη μας τι διοικητική δομή είναι, πόσο πιστή είναι στην κυβέρνηση. Μόλις έγινε πραξικόπημα Πόσες μονάδες έχουμε ακόμη εμπιστοσύνη ότι θα υποστηρίξουν την κυβέρνηση του Μαλή όταν ε, την υποστηρίζουμε εμείς ως Ένωση, ως γαλλικές στρατιωτικές δυνάμεις και αυτοί βέβαια οι δυνάμεις του Μαλή πρέπει να αναδιαρθρωθούν να, μπορέσουν να, να μπορέσουν να γίνουν έτοιμο πόλεμες. Βεβαίως ξέρουμε ότι αυτή τη στιγμή ε, στην πρώτη γραμμή της μάχης είναι η Λεγιώνα των Ξένων, η Γαλλική. Διάβασα ε, στο περιοδικό Spiegel, στην ηλεκτρονική του έκδοση, ότι οι δυνάμεις του Μαλή που συνεργάζονται με την ε, γαλλική εκστρατευτική δύναμη θανατώνουν τους ε, αντάρτες τους οποίους πιάνουν. Δεν είναι δυνατόν να συνεχιστεί αυτό. Άρα η κατάσταση απέχει πολύ από το να είναι ικανοποιητική. Άρα πρέπει να υπάρξει περισσότερη προσπάθεια από πλευράς μας, περισσότερη συμμετοχή. Δεν είναι δυνατόν ε, να θεωρήσουμε ότι αρκεί η Γαλλία να αναλάβει την ευθύνη όλων μας και άλλα ευρωπαϊκά κράτη πρέπει να συμβάλλουν περισσότερο. Δεν αρκούν ε, μεταγωγικά αεροσκάφη και διακήρυξεις. Και αυτό αφορά και τη δική μου κυβέρνηση. Αλλά θα ήθελα και η κάθε και τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα να εκφραστούν, να εκφράσουν αυτές τις προσδοκίες έναντι των κρατών μελών δημοσίως. Εκφραστείτε παρακαλώ δημοσίως, εκφράστε τις απαιτήσεις σας έναντι των κρατών μελών να δούμε λοιπόν τι θα κάνουν. Ευχαριστώ, Άντζου Νταφ. Κύριοι, μετά τα όσα είπε ο Μάικλ Γκάλαχαρ, συμμερίζομαι την ε, εντύπωση ότι υφιστάμεθα τώρα τις συνέπειες μια σημαντικής αποτυχίας στον τομέα των πληροφοριών. Νομίζω ότι εφησύχασαν και η Ένωση και οι Ηνωμένε Πολιτείε, ενώ σε ολόκληρο το Σαχέλ η κατάσταση επιδεινώνεται. Οπωσδήποτε, η υπηρεσία εξωτερικής δράσης δεν μας προειδοποίησε ότι η κατάσταση κατέρε τόσο ταχαίως. Ίσως να φταίω κι εγώ. Αλλά είχα την εντύπωση ότι η κοινή πεποίθηση ήταν ότι μπορούσε να ελεγχθεί η ε, πρόοδος των ε, Ισλαμιστών. Αλλά βλέποντας πώς εξεράγει η σύραξη στο Μαλίν... καθώς και την ε, τρομοκρατική επίθεση στην ε, Αλγερία, διαπιστώνω ότι ουδόλως ισχύει αυτό. Η κυρία Χίλαρη Κλίντον χθες παρουσίασε την κατάσταση έτσι ώστε κατέστησε σαφές ότι πρέπει να εμπλακούμε ουσιοδός και επιμακρών στην περιοχή. Θα ήθελα λοιπόν η Ένωση επίσης να επιβεβαιώσει αν συμφωνεί με αυτήν την εκτίμηση. Θεωρείται ότι πρέπει να προετοιμαστούμε για μια μεγάλη κλίμακος και μακροχρόνια και δαπανηρή πολιτική και στρατιωτική αποστολή σε όλη την έκταση του Σαχέλου. Συγκεκριμένα τώρα, η εκπαίδευση των στρατιωτικών ε, των Αφρικανικών χωρών. Εμείς μπορούμε να τους εκπαιδεύσουμε, αλλά πώς θα τους αποτρέψουμε από το να περάσουν μετά με την πλευρά των τζιχάντι. Γιατί ήδη είχαμε αρκετά τέτοια προηγούμενα. Πολλά. Διότι και στο Αφγανιστάν διαπιστώσαμε τέτοιες λιποταξίες. Εμείς εκπαιδεύαμε στρατιώτες, τους εξοπλίζαμε και μετά λιποτακτούσαν προς τους Ταλιμπάν. Εκπαιδεύαμε δηλαδή Ταλιμπάν. Όπως είπε και ο κύριος Ντόζο, αυτές οι ομάδες μάχης σε τι χρησιμεύουν αν δεν αναπτυχθούν εδώ και τώρα. Ποιες λοιπόν τέτοιες ομάδες μάχης μπορούμε να αναμένουμε ότι είναι σε θέση να αναπτυχθούν στο Σαχέλ ταχύτατα για να υποστηρίξουν τις ε, γαλλικές επιτόπου δυνάμεις. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ, Άντριου. Ήρθε εδώ ο Φρανσίς. Είναι εισηγήτρια για το ε, μέσο για τη σταθερότητα. Για τα χρηματοδοτικά θέματα έχετε ανακοινώσει 15 εκατομμύρια ευρώ ή 50 ότι θα δοθούν σε αυτήν την αποστολή. 50 εκατομμύρια. τις επόμενες δέκα μέρες το κόστος της γαλλικής επιχείρησης θα κοστίσει 30 εκατομμύρια ευρώ. Θα είναι δύσκολο ούτως ή άλλως να χρηματοδοτήσουμε αυτή την ε, προσπάθεια ατομικά το Η να χρηματοδοτησουμε αυτη την προσπαθεια ατομικα η αφορά το μέσο σταθερότητας. Ε, συζητήσαμε αρκετά το περασμένο φθινόπωρο, το φθινόπωρο του 12 δηλαδή, για το μέσο αυτό και σας είχα πει ότι υπάρχει ένα χρηματοδοτικό πρόγραμμα για το Βόρειο Μαλλί για την αναθεώρηση και συγχρονισμό του τομέα της ασφάλειας για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας γενικά στο Σαχέρι. Ε, υπήρχε όμως ένα πρόβλημα. Ε, καλό είναι να υπάρχουν προγράμματα για το Σαχέλ. Θα ήθελα να μου πείτε τι μπορούμε να διδαχθούμε τελικά από όλα αυτά τα προγράμματα τι λειτουργήσε, τι πήγε καλά, τι δεν πήγε καλά στο Βορρά. Είναι σημαντικό να δούμε με ποιους δουλέψαμε, τι συνέβη με αυτούς που συνεργαστήκαμε, σήμερα με ποιους είναι. Έχουμε επαφή μαζί τους. Θα πρέπει να υπάρχει μία συνέχεια νομίζω. Και το δεύτερο που θέλω να πω είναι ότι ακούγονται ψήθυροι ότι θα γίνει μία ειρηνευτική διάσκεψη ε, στον ΟΗΕ υπό την αιγίδα του Πρόντι, με... που θα συμμετάσχουν και οι περιφερειακές δυνάμεις. Και όλοι οι φορείς που είναι έτοιμοι να συμμετάσχουν και σε περιφερειακό επίπεδο, από το βορρά, από το νότο, θα συμμετάσχουν σε αυτή τη διάσκεψη. Η Ευρωπαϊκή Ένωση στηρίζει αυτή την ιδέα, την προωθεί. Τελευταίο σημείο για τις ομάδες μάχης που ακούστηκαν πολλές φορές το προηγουμένως, στη Γερμανία κάνουμε, κάνουμε μια συζήτηση ότι εμείς δεν μπορούμε να παρέμβουμε στο Βόρειο Μαλί, δεν έχουμε τα ελικόπτερα. η δοκιμία έγινε στο Αφγανιστάν. Μου λέγανε ότι... Μου είπαν όμως ότι αν υπήρχαν αυτές οι ομάδες μάχης, οι Γερμανοί θα μπορούσαν να συμμετάσχουν. μου είχαν πει ότι υπήρχε πρόβλημα με τα γερμανικά ελικόπτερα. Τουλάχιστον αυτό συζητάνε στο Bundestag. Ε, εάν υπήρχαν οι ομάδες μάχης διαθέσιμες, δεν θα είχαμε πρόβλημα. Η κυρία Κιλ Νίλσον. Ευχαριστώ. Να κάνω κάποια ερωτήματα που θέτει η ομάδα των Πρασίνων. Καταρχάς, έχει νόημα να ξεκινήσουμε μια εκπαιδευτική αποστολή τη στιγμή που οι περισσότεροι στρατιωτικοί ε, δραστηριοποιούνται στο μέτωπο. Το δεύτερο, το είπε και ο συνάδελφος, τον, το πρόβλημα των λιποταξιών, που είναι σημαντικό. Είχαμε την ίδια εμπειρία. Ε, εκπαιδεύσαμε στρατιωτικούς στη Σομαλία και είδαμε ότι αυτοί που εκπαιδεύσαμε συνεχεία λιποτακτούσαν στις ε, ομάδες Σαμπάπ. Επίσης, οι μονάδες που εκπαίδευσαν οι στο βόρειο Μαλί, εν μέρη μπήκαν στο αντάρτικο των Αρέγ. τρεις μονάδες και ορισμένοι συμμετείχαν ε, στις 22 Μαρτίου στο πραξικόπημα. Δεν υπάρχει κίνδυνος λοιπόν να εκπαιδεύσουμε ανθρώπους ε, οι οποίοι μετά τι θα, κάνουν αυτή την ε, γνώση. Θα προωθήσουν άλλα συμφέροντα, Επίση, δεν αμφισβητούμε βέβαια την νομιμότητα τη γαλλική παρέμβαση, αλλά είναι νόμιμο και θεμητό να παρεμβαίνουμε για να εκπαιδεύσουμε ένα στρατό όταν δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή τουλάχιστον δημοκρατική διαδικασία στη χώρα. Είναι θεμητό επί της αρχής να εκπαιδεύουμε στρατιωτικούς τη στιγμή που δεν υπάρχει μια πολιτική διαδικασία που εξασφαλίζει τον έλεγχο αυτών των στρατιωτικών. Είναι ένα θέμα άλλο που θέτουν οι πράσινοι. Τελευταίο ερώτημα για τον κύριο Westcott. Αληθεύει ότι οι Υπουργοί Εξωτερικών έχουν απελευθερώσει 230 εκατομμύρια ευρώ. Ή μάλλον, να το πω πιο σωστά. Τα 230 εκατομμύρια ευρώ που προβλέπονταν ε, για την περιοχή μπορούν να χρησιμοποιηθούν τώρα για την αναπτυξιακή βοήθεια. Αφορά τον έλεγχο του χρήματος. Σε ποιον δίνουμε τον έλεγχο αυτού το, αυτών των χρημάτων. Σε μία μη νόμιμη κυβέρνηση. Επίσης, για μας τους οικολόγους, πιστεύουμε ότι η φτώχεια στο Μαλί προκύπτει από την κακή χρήψη εν μέρη των σημαντικών του σημαντικού πλούτου από το φυσικό αέριο και από τα μεταλλεύματα και ορυκτά που έχει το Μαλί. Υπάρχει ένα μονοπόλιο, υπάρχουν μεγάλες ε, ε, πολυεθνικές, η Ρέβα του Νίγηρα έχουν τον έλεγχο αυτών των ε, φυσικών πόρων και τα λεφτά πηγαίνουν σε κάποιους διεφθαρμένους πολιτικούς. Εμείς ως Ευρωπαϊκή Ένωση, ποια αναπτυξιακή βοήθεια βιώσιμη προωθούμε για τη Σαχέλ με ποια συμμετοχή. Πώς εξασφαλίζουμε τη δικαιοσύνη στον, στην κατανομή του πλούτου της περιοχής. Για τη Γαλλία, ο Υπουργός Ανάπτυξης, ο Πασκάλ Κανθα, είναι ένας παλιός ευρωβουλευτής, τον ξέρουμε. Δουλεύει αυτή τη στιγμή, ούτω ώστε να δούμε τι θα κάνουμε ε, μετά το τέλος της κρίσης στο τομέα της ανάπτυξης. Αυτό το κάνει η Γαλλία. Η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να συνεισφέρει σε αυτή την προσπάθεια ανάπτυξη, βιώσιμης ανάπτυξης του Σαχέλ. Ευχαριστώ που ακούσατε όλες αυτέ τι ερωτήσει και που θα απαντήσετε. Ευχαριστώ. Ο κύριος Λίζεκ. Ευχαριστώ. Ακούσαμε πολλά για τη στρατιωτική παρέμβαση. Εσείς που είσαστε ειδικοί, κύριοι, τι πιστεύετε για την πολιτική κατάσταση στο Μαλί. Ξέρουμε ότι το Μαλί Ξέρουμε ότι δεν είναι μια δημοκρατική οργα, ε, χώρα που λαμβάνουν χώρα, σφιγμομετρήσεις όπως στην Ευρωπαϊκή Ένωση ή στην, ε, στις Αλλά τι πιστεύετε ότι ο, λαός του Μαλή, ο πληθυσμό του Μαλή πιστεύει για τη γαλλική παρέμβαση. Επίσης, πώς, πώς υποστηρίζει ο λαός του Μαλή την κυβέρνηση. Αν φύγουν οι Γάλλοι στρατιωτικοί, θα καταρρεύσει πάρα αυτά η κυβέρνηση του Μαλή. Ο λαός του Μαλή υποστηρίζει αυτή την κυβέρνηση ή βασίζεται απλώς στην γαλλική στρατιωτική παρουσία αυτή η κυβέρνηση. Ο κύριος Λανσμπέργκης. Υπάρχει περίπτωση να κλιμακωθεί ο πόλεμος της Αλ-Κάιντα στο Μαλί. Δεν ξέρουμε τις προθέσεις της Αλ-Κάιντα Τι έχουμε προβλέψει στο σενάριο που η Αλ-Κάιντα προκαλέσει ευρύς πολέμους στην Αφρική αν κάνει επιθέσεις ε, στην ε, Ευρώπη. Τι θα κάνουμε. Η Γαλλία θα ζητήσει βοήθεια από το ΝΑΤΟ. Υπάρχει ενδιαφέρον να εμπλακεί το ΝΑΤΟ και οι Ηνωμένε Πολιτείε σε έναν μαύρο αφρικανικό πόλεμο. Τι πιστεύει η Γαλλία. Η Γαλλία που είναι στην πρωτοκαθεδρία τώρα αυτών των προσπαθειών είναι έτοιμη να αναλάβει και να απαντήσει σε μια τέτοια πρόκληση. Σας ευχαριστώ που μας ενημερώνετε, Λέω ο κύριος Κέλαμ. Η ευρωπαϊκή παρέμβαση στο Μαλί ήταν μια απλή αντίδραση σε τρομοκρατικέ δραστηριότητε, Μια καθυστερημένη μάλιστα αντίδραση, όπως είπαν οι συναδελφοί μου. Πρέπει όμως να μην ξεχνάμε ποιο είναι το ευρύτερο πλαίσιο. Είναι σαφές πλέον ότι θα χρειαστούμε μια μακροπρόθεσμη στρατηγική από πλευράς Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη Σαχέλ η περιοχή αυτή είναι πολύ πιο κοντά από το Αφγανιστάν σε εμά. Και οικονομικά και στρατηγικά μα ενδιαφέρει πολύ περισσότερο. Πρέπει να είμαστε προετοιμασμένοι για τις όποιες εξελίξεις. Και σε πολιτικό επίπεδο. Τι θα κάνουμε με τις γειτονικέ χώρες, με την Αίγυπτο, της οποίας ο πρόεδρος ονόμασε αυτή την παρέμβαση επίθεση ή την Τινησία θα είπε ότι δεν θα πρέπει οι Ευρωπαίοι να παρέμβουν. Μόνο οι Αφρικανοί θα πρέπει να επιλύσουν αυτή την κρίση. Αυτή η παρέμβαση των Γάλλων ή της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν αντιμετωπίζει τα αίτια του προβλήματος, που είναι η τρομοκρατία. Στην νοτιοανατολική Λιβύη ε, γίνεται εκπαίδευση τρομοκρατών που έρχονται από το Αφγανιστάν και που τους αποστέλνουν συνεχεία στο Μαλί. Πρέπει να αντιμετωπίσουμε όλα αυτά τα ερωτήματα. Ε, το τρίτο πρόβλημα αφορά την εσωτερική κατάσταση του Μαλί. Νομίζω ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να βοηθήσει για να ενισχυθεί η εσωτερική σταθερότητα του Μαλί. Από ό,τι φαίνεται, ο πληθυσμός πλέον ε, λαμβάνει τη βοήθειά μας και είναι σαφές ότι τα εξτρεμιστικά στοιχεία είναι η μειονότητα. Αλλά θα πρέπει να δώσουμε μεγαλύτερη οικονομική βοήθεια για μεγαλύτερη κοινωνική δικαιοσύνη. Το ηθικό δίδαγμα είναι ότι μια και ξεκινήσαμε αυτή την επιχείρηση, δεν μπορούμε να σταματήσουμε στα μισά. Χρειαζόμαστε μια πακροπρόθεσμη στρατηγική. τέθηκε το ερώτημα για τις ομάδες μάχης. Θέλω και εγώ να μου δώσετε μια απάντηση. Ο Τζολ Στάνο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ζητώ συγγνώμη που δεν ήμουν εδώ νωρίτερα. Ε, υπάρχει πάντοτε σύγκρουση μαζί με τις διάφορες επιτροπές όπου γίνονται διάφορες ενδιαφέρουσες συζητήσει, όπως η κατάργηση της θανατική ποινή στην Ταϊβάν, ε, στην ε, ε, μιλήσαμε ήδη για το Αμαλή, μιλάσαμε για τις εμπειρίες στο κέρας της Αφρικής και στην Ουγγάντα, όπου έγινε μια εκπαιδευτική αποστολή για τον Σομαλικό στρατό και υπήρξε πρόβλημα ε, λιποταξιών, αυτομολύσεων, δηλαδή χρήση χρημάτων ε, της Ευρωπαϊκής Ένωσης για εκπαίδευση στρατιωτικών, οι οποίοι μετά έφευγαν και πήγαιναν στην Ισομπάμπα. Στο BBC έγινε σχετική αναφορά για το Βόρειο Μαλίο που ισχυρίστηκε ο δημοσιογράφος ότι σημαντικές, ε, ε, σημαντικό τμήμα των ε, ανταρτών ήταν πριν στρατιώτες του στρατού της χώρας. Πώς θα αποφύγουμε λοιπόν τα ίδια προβλήματα που είχαμε στην Ουγγάντα, δηλαδή να εκπαιδεύουμε τους στρατιώτες του Μαλί με χρήματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και μετά αυτοί τελικά να πηγαίνουν με τους αντάρτες. Πώς θα τα αποφύγουμε αυτό. Ευχαριστώ. Πριν να δώσω το λόγο στους προσκεκλημένους μας, να δώσω ε, κάποιες παρατηρήσεις, να κάνω κάποιες παρατηρήσεις. Αυτή η θέμα της ε, λιποταξίας, αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Έχει γίνει Έχει γίνει αυτό και στη Σομαλία γιατί από τα τρία σώματα που εκπαιδεύτηκαν από την αποστολή μας στη Σομαλία είδαμε ε, λιποταξίες που όμως δεν πήγαν προς τους Σεμπάμπ. Ήταν άνθρωποι οι οποίοι εκπαιδεύτηκαν και μετά πήγαν στα ε, χωριά τους χωρίς να συμμετέχουν στις μάχες. Εντάξει, υπήρξαν κάποια αλλά σίγουρα όχι στις αναλογίες που κάποιες φορές αφήνουμε να εννοηθεί. Προσοχή λοιπόν, αν και είναι ζήτημα για τη συνέχεια, που μάλιστα μπορεί να συνδεθεί και με το θέμα των ε, απαιτήσεων και των ε, αποχωρήσεων από το στρατό του Μαλή, των ε, που είναι και αυτό το θέμα που μας απασχολεί σήμερα. Έπειτα, μπορείτε να μας επιβεβαιώσετε αυτό που μας είπαν χτες, ότι δηλαδή το θέμα του Μαλή δεν συζητήθηκε καθόλου στο, Μαλή, στο ΝΑΤΟ, με συγχωρείτε, και ότι εν μέρη για ένα λόγο ενός κόμματος της, ε, συγγνώμη, μιας αντιπολίτευσης τουρκικής η οποία δεν δέχεται να αποκαλούνται Ισλαμιστές οι ομάδες των ανταρτών κατά των οποίων ε, γίνεται ο πόλεμος αυτή τη στιγμή. Όλοι γνωρίζουμε δε τώρα ότι είναι πολύ σημαντικό και ότι η στρατιωτική αυτή επιχείρηση δεν θα έχει κανένα νόημα εάν δεν συνοδευτεί και από πολιτικό, πολιτική διαδικασία. Ποιοι είναι οι συνομιλητέ που έχει η Ευρωπαϊκή Ένωση λοιπόν σε πολιτικό επίπεδο. Συζητάει η Ευρωπαϊκή Ένωση με το MNLA που έχει αποστασιοποιηθεί από τις Ισλαμικές ομάδες και έπειτα καταλάβαμε ότι υπάρχει μια, ένας διχασμός ε, στο Ανσαρτίν με ένα κομμάτι της ομάδας το οποίο αφήνει τις ε, πόλεμες δράσεις για να μπει στις διαπραγματεύσεις. Καταλαβαίνω ότι θα είναι κάποιο αρχικό στάδιο αξιολόγηση αυτό, αλλά εν πάση περιπτώσει ποιοι είναι οι συνομιλητέ που έχει τώρα η Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν μιλώ για τα κρατημέλη. Ξέρω πω κάποια κρατημέλη έχουν επαφέ με την τάδε την ομάδα, αλλά από τη δική μα πλευρά τη Ένωση, ποιοι είναι οι συνομιλητέ μα για να συνοδευτεί αυτή η κατάσταση από πολιτική διαπραγμάτευση. Πολλά, πολλά ερωτήματα λοιπόν έχουν τεθεί. Ο Νίκολας Βέσκοτ να απαντήσει πρώτα. Ναι, ευχαριστώ Πρόεδρε. Πολύ σημαντικά ερωτήματα και θα προσπαθήσω να απαντήσω σε όσα μπορώ και σε κάποιο βαθμό συλλογικά. Τόσο ο κύριος Γκάλερ όσο και ο κύριος Νταφ ρώτησαν τη στρατηγική μας προσέγγιση και τις προβλέψεις. Κοιτάξτε, δεν ήταν κεραυνός εν εθρία. Γνωρίζαμε και το γνωρίζαμε εδώ και πολύ καιρό πως ε, το Σαχέλ είναι μια εξαιρετικά ευάλωτη ε, και ζώνη γεμάτη διακοιμάνσεις. Υπήρχε σχετική στρατηγική. Ήταν ένα μακροπρόθεσμο πρόβλημα που χρειαζόταν μια μακροπρόθεσμη λύση. Ακόμα σε αυτό είμαστε δεσμευμένοι, σε μακρόπνοη λύση και όχι μόνο στο να ξεπεράσουμε την άμεση κρίση. Γιατί διαφορετικά θα κάνουμε συνέχεια τα ίδια πράγματα. Έχουμε ότι είναι διάφορα τα στρατεύματα, διάφορες ομάδες, ξέρουμε ότι πιέζονται ιδεολογικά, ξέρουμε ότι υπάρχουν εγκληματικές δραστηριότητες που για αιώνες αναπτύσσονται σε αυτές τις περιοχές, λαθρεμπόριο, τσιγάρων, όπλων, ανθρώπων, ναρκωτικών. Ε, το πρόβλημα λοιπόν είναι γνωστό. Τώρα, αυτό που συνέβη τον Ιανουάριο φέτος ήταν μια ακραία επιτάχυνση. Και έτσι δύο πράγματα κατέστησαν σαφή. Πρώτον, ότι οι αντάρτες, ε, οι Ισλαμιστές τζιχάντι είχαν αποφασίσει να καταλάβουν όσο γίνεται περισσότερο, περισσότερα εδάφη και να τα ελέγξουν. Ε, ε, αυτό δεν είχε γίνει πέρυσι και μάλιστα θέλησαν να ενεργήσουν πριν να προετοιμαστεί η διεθνής κοινότητα για να μπορέσουν να ανακτήσουν τον έλεγχο του Νουπορά. Έπειτα κατέστησε σαφέ πως ο Μαλνέζικο στρατό ο ίδιο, αν και είχε πει ότι μπορούσε να τα βγάλει πέρα, δεν μπόρεσε να σταματήσει του τρομοκράτε. Και η κυβέρνηση του Μαλή ζήτησε από το ΝΟΙΕ και από την Ευρωπαϊκή Ένωση βοήθεια. Η προσωρινή κυβέρνηση, ο πρόεδρο Στραωρή είναι η πιο νόμιμη κυβέρνηση που έχουν. Εν πάση περιπτώσει, έχει πάρει τη θέση του, έχει ορκιστεί στο Σύνταγμα κτλ. Ήταν η νόμιμη αρχή λοιπόν που έκανε αυτή την έκκληση και οι Γάλλοι ήταν σε θέση να ανταποκριθούν και το έκαναν. Γιατί εμεί δεν ενεργήσαμε νωρίτερα. Είχαμε ήδη υποδείξει ποια στοιχεία ήταν απαραίτητα για την λύση. Και εμείς συνεργαζόμαστε με τους Αφρικανούς εταίρους μας για να τα υλοποιήσουμε όλα αυτά. Τώρα τα όσα έγιναν τον Ιανουάριο επιτάχυναν όλη αυτή τη διαδικασία ώστε χωρίς ε, στρατιωτική παρέμβαση, επέμβαση θα είχε επιδεινωθεί πολύ τα, η κατάσταση και υπήρχε μεγάλος κίνδυνος οι αντάρτες να καταλάβουν ολόκληρο το κράτος του Μαλή με καταστροφικές επιπτώσεις για τον ίδιο τον λαό της χώρας. Οπότε συνεχίζουμε και προσπαθούμε να επιταχύνουμε συλλογικές λύσεις. Εμείς θέλουμε μια αφρικανική λύση για το αφρικανικό αυτό πρόβλημα. Ωστόσο, αυτή τη στιγμή ο λαός του Μαλή ζήτησε την επέμβαση της διεθνούς κοινότητας και εμείς ως Ευρωπαϊκή Ένωση, η Γαλλία και άλλα μπορούν να βοηθήσουν. Είναι λοιπόν προς το συμφέρον μας αλλά και προς το δικό τους τελικά η τελική λύση να είναι μια νόμιμη, δυνατή, δημοκρατικά εκλεγμένη κυβέρνηση στο Μαλί με αντίστοιχη κρατική δομή που θα μπορεί να επιβάλλει το κράτος δικαίου από πλευράς αυτής της νόμιμης κυβέρνησης. Αυτός είναι ο απότερος στόχος. και ε, καταρχήν πρέπει να σταθεροποιηθεί η κατάσταση. Αυτό πρέπει, θέλει να κάνει η Γαλλία, προσπαθεί να το κάνει, να εκπαιδεύσει τον στρατό του Μαλή, όχι μόνο ώστε να μπορεί να είναι αποτελεσματικός, αλλά και νόμιμος, νομότυπος που θα ενεργεί με βάση τον ανθρωπιστικό νόμο. Μπορεί να μην συμβαίνει ακόμα, αλλά η επιμονή μας σε αυτό το πολιτικό οδικό χάρτη και πολιτική διαδικασία που θα συμπεριλαμβάνει και εκπροσώπους των ομάδων στο Βορρά, οι πολλοί από τους οποίους έχουν εξοριστεί στον Νότο, γιατί αν βρίσκονταν στο Βορρά κινδυνεύει η ζωή τους. Λοιπόν, θέλουμε να βρεθεί μια πολιτική καθολική λύση. Έτσι, η εκπαίδευση για το στρατό σημαίνει εκπαίδευση στον ανθρωπιστικό νόμο, στη ε, ε, εκδημοκρατισμό κτλ. Αλλά όλα αυτά, όπως καταλαβαίνετε, δεν γίνονται εν μία νυχτή. Δεν υπάρχει μαγικό ραβδί. Η εκπαίδευση λοιπόν του Μαλνέζικου στρατού αλλά και των στατευμάτων της αφίσμα που θα, που, που θα επέμβουν είναι ένα βασικό στοιχείο για να εξασφαλίσουμε την αποτελεσματικότητα αυτής της διαδικασίας. Επίσης, ε, ποιος θα είναι επικεφαλής. Διοίκηση και έλεγχος. Ποιος θα είναι επικεφαλής, δεν έχουμε απάντηση για την ώρα. Αυτή είναι όμως η πιο σημαντική ερώτηση που θα ρωτήσουμε. Στις 29 Ιανουαρίου χρειάζεται να υπάρχει σαφής και αποτελεσματική διοικητική δομή, διότι έρχονται στρατεύματα από διάφορες πλευρές ε, και πρέπει να συνεργαστούν. Διαφορετικά δεν θα επιτύχουμε. Υπάρχουν ερωτήματα λοιπόν που δεν μπορούμε να απαντήσουμε για την ώρα αλλά ξέρουμε ότι πρέπει να τα απαντήσουμε αν θέλουμε η επιχείρηση αυτή να είναι επιτυχής. Επόμενο ερώτημα. Προγράμματα για την ασφάλεια στον Βορρά. Πολύ θα θέλαμε να το εφαρμόσουμε αυτό όσο γίνεται. Έχουμε εντοπίσει ποιοι είναι οι μάρτυρες η ίδια η κυβέρνηση με, υπό τον πρώην πρόεδρο είχαν, είχε φτιάξει το PSBN, δεν θυμάμαι ποιο ήταν ο, ολόκληρος ο τίτλος, για την ε, εγκαθίδρυση της ασφάλειας και της κυβέρνησης στην, στον βορρά της χώρας. Αλλά δυστυχώς ε, ελάχιστα έγιναν και πολύ αργά και όχι με την αποφασιστικότητα που ήταν απαραίτητη. Το συγκεκριμένο πρόγραμμα λοιπόν αυτή τη στιγμή ε, είναι σε αναστολή. Μπορούμε να αναδιπλώσουμε τα χρήματα και να τα χρησιμοποιήσουμε από τη στιγμή που θα είναι χρήσιμο να τα κάνουμε κάνουμε. Και μιλάμε για τα προγράμματα σταθερότητας, τα οποία μπορούν πολύ γρήγορα να φέρουν επιχειρησιακή στήριξη στην κυβέρνηση του Μαλή η οποία είναι απαραίτητη. Και αυτό θα είναι τμήμα τη αποστολή αξιολόγηση των αναγκών που σα περιέγραψα στην αρχή. Θα είναι μια υπηρεσιακή αποστολή που θα δει όχι μόνο τι εξελίξει, του αναπτυξιακού στόχου, αλλά και τι άμεσε δραστηριότητε. Τώρα, για την ε, αναπτυξιακή βοήθεια. Να σας δώσω την, θα σας αφήσω την Επιτροπή Ανάπτυξης να σας δώσει όλες τις λεπτομέρειες, αλλά όταν έγινε το πραξικόπημα πέρυσι, αναστήλαμε όλη τη βοήθεια που δίναμε άμεσα στην κυβέρνηση του Μαλή, γιατί δεν υπήρχε κανένας υπεύθυνο για το τι θα κάνανε αυτά τα χρήματα. Συνεχίσαμε να στηρίζουμε την άμεση βοήθεια προς τον λαό, εκείνη δηλαδή που δεν περνούσε από την κυβέρνηση. Και είμαστε μέσα στο ίδια διαδικασία υπό το 10ο EDF, ε, αναπτυξιακό πρόγραμμα, ε, και έτσι έχουμε καταλήξει σε περίπου 90 εκατομμύρια ευρώ τα οποία πάγωσαν και 150 ακόμη ε, για στήριξη προγραμμάτων τα οποία όμως δεν έχουν ακόμα δεσμευτεί. Τώρα αυτά τα νούμερα που σας λέω θα έπρεπε να τα επιβεβαιώσει και η Επιτροπή Ανάπτυξης αλλά γι' αυτό τον λόγο είναι τόσο σημαντικό να δούμε τώρα τι μπορούμε να κάνουμε με αυτά τα χρήματα που να είναι χρήσιμο, γιατί ο λαός του Μαλή έχει απελπιστικές ανάγκες. Μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε την κυβέρνηση ως μέσο. Μπορούμε να ελπίσουμε σε ανοικοδόμηση από τη στιγμή που θα υπάρχει νόμιμη κυβέρνηση. Ποιε είναι οι πιο επίγουσες ανάγκες και πού μπορούν να δαπανηθούν ικανοποιητικά και αποτελεσματικά αυτά τα χρήματα. Δεν ξέρουμε ακόμα τις απαντήσεις εάν δεν πάμε επί τόπου να δούμε τι γίνεται. Αυτή είναι η προτεραιότητα και μετά θα επανέλθουμε με πληρέστερε απαντήσεις για το πώς θα χρησιμοποιήσουμε αυτά τα Πολιτική κατάσταση τώρα που έχει ε, θίξει ο κύριος Λίζεκ. Όλες οι αναφορές που άκουσα υποδεικνύουν ότι ο λαός του Μαλή είναι εξαιρετικά ευγνώμονας για την παρέμβαση της Γαλλίας. Είμαι βέβαιος ότι πολλοί δημοσιογράφοι ψάχνουν να βρουν κάποιον που θα επικρίνει την γαλλική επέμβαση. Δεν έχουν βρει ακόμα κανέναν μέσα στη χώρα, αλλά, μπας περιπτώσει, όλοι συνειδητοποιούν ότι χωρίς την παρέμβαση αυτή οι αντάρτε θα είχαν φτάσει στην Μπαμακό αυτή τη στιγμή. Είναι εξαιρετικά καλά οπλισμένοι, πολύ καλά εκπαιδευμένοι και αποφασισμένοι και είναι και ε, πραγματικά αμήλικτοι. Το είδαμε από τη συμπεριφορά του στο Βορρά. Υπάρχουν, έχουν και χρήματα από τις ομοιρίες διαφόρων, αλλά τα χρήματα νομίζω προέρχονται από εγκληματικές ε, δραστηριότητες, κυρίως λαθρεμπόρια ναρκωτικών και όπλων. Και αυτό γεμίζει τις τσέπες του σταθερά. Γι' αυτό και τα προβλήματα του Μαλή δεν μπορούν να λυθούν μόνο μέσω του Μαλή. Είναι περιφερειακό το πρόβλημα, συμπεριλαμβανομένης του λαθρεμπορίου ναρκωτικών σε ολόκληρη τη Δυτική Αφρική. Και αυτό κοιτάμε αυτή τη στιγμή με την επίδεση εξωτερικής δράσης. Το, η, στρατηγική για το Σεχέλ παραμένει. Η στρατηγική για το Σεχέλ και είναι εξαιρετικά σημαντικό να στηρίξουμε το Μαλί, τη Μαυρετανία, το, την Πουργίνα Φάσο, ώστε να μην υπάρξει αυτός, αυτή η μετάδοση κίνδυνος μετάδοση. Το είδαμε ήδη στην Αλγερία με την τραγωδία στην εγκατάσταση ε, του φυσικού αερίου. Η Σαχάρα είναι λίγο σαν τη θάλασσα, δεν έχει ξεκάθαρα σύνορα εκεί. Εάν κανείς είναι ευκίνητος μπορεί να ε, ε, πάει από τη μια χώρα στην άλλη στο φύ. Πρέπει να ενισχυθεί και η Νιγηρία, η Νιαμέη. Είναι και αυτό το τμήμα της στρατηγικής μας. Πολύ κίνδυνοι, κίνδυνοι δρομεροί. Ε, οι αυτή είναι Σαφή. Επηρεάζεται λοιπόν ολόκληρη η περιφέρεια και γι' αυτό η δικιά μας επιχείρηση θα είναι επιτυχής μόνο εάν συνεργαστούμε με την ΕΚΟΒΟΣ και με την Αφρικανική Ένωση. Και αυτό είναι ο στόχο τη επόμενη μα επαφέ, ότι δηλαδή να είμαστε κομμάτι των διεθνών συλλογικών προσπαθειών στη στήριξη του μαλινέζικου λαού. Σας ευχαριστώ. Καταρχήν για το θέμα του ΝΑΤΟ και του ρόλου του ΝΑΤΟ στο Μαλί. Νομίζω ότι καλύτερα να ρωτήσετε στους εκπροσώπους του ΝΑΤΟ για το θέμα αυτό. Όπως και εγώ παρακολουθώ τις συζητήσεις που γίνονται για αυτόν. Προς τον κύριο Τάνοκ. Κάτι συμπληρωματικό για τις προσπάθειές μας στην Σομαλία γιατί είπατε ότι υπήρξαν κάποιες ε, λιποταξίες. Βεβαίως, ε, βεβαίως ε, παλιά όταν στείλαμε πίσω τους 500 900 στρατιώτες που τους είχαμε πάρει από την περιοχή τους, τους, πήραμε, τους πήγαμε στον Μπιχάγκα. Είχε να κάνει με την κατάσταση ασφαλής Σομαλία, γι' αυτό χρειάστηκε να τους βγάλουμε από τη Σομαλία τους πήραμε λοιπόν και πήραμε λοιπόν άτομα από διάφορες περιοχές της χώρας και τους ε, ε, βάλαμε σε ένα τάγμα. Δημιούργησε πολύ ισχυρή, ε, ισχυρό πνεύμα μονάδας. Τους βοήθησε μετά. Όταν τους στείλαμε πίσω στη χώρα του, ε, ορισμένοι απλώς γύρισαν στις οικογένειές τους γιατί έλειπαν έξι μήνες. Αλλά πρέπει να πω ότι περισσότεροι μετά επέστρεψαν. Μέχρι στιγμής έχουμε εκπαιδεύσει 3.000. Όλοι πήγαν στην πρώτη γραμμή του μετόπου, πολέμησαν πολύ καλά. Υπήρξαν μερικές λιποταξίες, αλλά όπως σας είπα το ποσοστό είναι 10%. Ξέρετε, ακόμη και στο Βαλγικό στρατό, όταν προσλαμβάνονται στρατιώτες, κάποιοι μετά εγκαταλείπουν. Δεν ξέρω τι έγινε στο Βρετανικό στρατό. Α, μάλιστα, μάλιστα. 3% το ποσοστό, μάλιστα. Κοιτάξτε, αλλά πρέπει να επαναλάβω ότι τους είδα αυτούς τους στρατιώτες. Ήταν ε, ιδιαίτερα έτοιμο πόλεμοι. Ο Λίν Πάσκο, ο βοηθός γενικός γραμματέας των ΗΠΑ, μας είπε ότι οι στρατιωτικές δυνάμεις που εκαδεύσατε έπαιξαν ε, καταλητικό ρόλο στα πλαίσια των ε, αφρικανικών δυνάμεων γενικότερα. Μέχρι τότε απλώς έλεγαν μερικούς δρόμους στατικά στο Μογκαντήσου αλλά αυτοί οι 3.000 άνδρες πήγαν με τις ε, δυνάμεις ε, του Amazon στην πρώτη γραμμή και έχουν ανακατακτήσει το μεγαλύτερο τμήμα της επικράτειας της Σομαλίας από την Al-Shabaab. Και τώρα βλέπουμε λιποταξίες από την Al-Shabaab προς τις δυνάμεις του Σομαλικού στρατού και ε, προσπαθούμε τώρα να τους εντάξουμε στις δικές μας στρατιωτικές δυνάμεις. Βέβαια είμαστε στην άλλη πλευρά τώρα τη Αφρική σε σχέση με το Μαλί τώρα για τις ομάδες μάχης. Βέβαια σημαντική ερώτηση. Η εύκολη απάντηση θα ήταν μα δεν υποβλήθηκε έτοιμα ούτε από το Μαλί, ούτε από τους Γάλλους, ούτε από τη διεθνή κοινότητα. Αλλά το έχουμε υπόψη μας, ε, προγραμματίζουμε γι' αυτό. Θα είμαι ειλικρινή. Οι δυνάμει αυτές, τίθεται το ερώτημα, έχουν αξιοποιηθεί όσο ε, θα μπορούσαν. Πρέπει να είμαστε ειλικρινεί λοιπόν. Οι μόνε δυνάμει που μπορούσαν να αξιοποιηθούν ήταν οι γαλλικέ δυνάμει. Γιατί ήταν ήδη στην περιοχή. Ακόμη και οι Αμερικανοί χρειάζονταν κάποιο χρόνο. Αναπτύχθηκαν λοιπόν σύντομα γιατί ήταν εκεί και τώρα στέλνουν δυνάμει από τη Γαλλία. Υπάρχει μια άλλη ομάδα μάχη που αποτελείται από γαλλικέ, γερμανικέ και πολωνικέ δυνάμει. Η γαλλική επιχείρηση είχε όπως ξέρετε πολύ καλά, άμεσα αποτελέσματα. Υποστηρίχθηκε από διάφορες χώρες μέλη, από τη διεθνή κοινότητα. Δεν υπάρχει ευρωπαϊκή σημαία, εντάξει. Αλλά είναι τμήμα της ευρωπαϊκής αντιμετώπισης του θέματος. Εν παρόδο υπενθυμίζω το άρθρο 44 της συνθήκης όπου λέει ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση ε, μπορεί να παρακαλέσει ένα ή περισσότερα κράτη-μέλη να δράσουν εξ ονόματός της στα πλαίσια του τομέα άμυνας και ασφάλειας. Δεν θέλουμε να περιοριστούμε σε αυτό, αλλά post factum μπορεί να ενταχθεί στην εφαρμογή αυτού του άρθρου. Τελείωσε ο ρόλο λοιπόν ε, των ομάδων μάχης. Ορισμένοι είπατε ότι θα πρέπει μακροπρόθεσμα να ασχοληθούμε με το θέμα αυτό. Θα υπάρξει και μια φάση σταθεροποίηση. Ξέρω ότι το σκέφτονται και στο Ρωμένα Έθνη και εμεί το σκέφτομαι. Είμαι υπέρ τη ομάδα μάχη. Θα υπάρξει χρήση ομάδα μάχη. Πιθανώ. Ένα ευρύτερο θέμα. Σε τι χρησιμεύουν οι ομάδε μάχη. Οπωσδήποτε θα συζητηθεί στο Δουβλίνο στη συνάντηση των διευθυντών ασφάλειας και άμυνας θα το συζητήσουμε προετοιμάζοντας το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, όπου η άμυνα φέτος το Δεκέμβρη θα είναι θέμα στην ημερήσια διάταξη. Το θεμελιώδες όμως ερώτημα που θα θέσουμε στα κράτη-μέλη είναι, ανάλογα βέβαια τι θέλουν να κάνουν και τα κράτη-μέλη, τα... οι ομάδες μάχης είναι μέσο για την ε, κατανομή καθηκόντων ή είναι μέσο μάχης. Υπάρχουν πολλέ ε, προτάσει. Για παράδειγμα, θα μπορούσε να υπάρχει ένα, ε, η ιδέα κάποιο κράτος να αναλαμβάνει τον ε, ε, ηγετικό ρόλο. Ξέρουμε ότι οι μεγαλύτερες χώρες θα μπορούσαν να παίξουν μεγαλύτερο ρόλο, αλλά ακόμη το εξετάζουν οι χώρες μέλη. Θα είναι λοιπόν στις προσεχείς ημερήσεις διατάξεις μας, αλλά εξαρτώμεθα από τις προθέσεις των κρατών μελών. Σε τι κατάσταση τώρα είναι ο στρατός του Μαλή. Έχουμε εικόνα γι' αυτό, καλή εικόνα. Υπήρξε γαλλική αποστολή που εξέτασε το θέμα αυτό. Υπάρχουν κάποιες μονάδες που είναι πολύ καλές, κάποια τάγματα. Υπάρχουν και κάποιες, ε, υπάρχει μάλιστα και ένα τάγμα του Αρέγ, το οποίο σταθμεύει στο βορρά. Οι Αμερικανοί έχουν εκπαιδεύσει κάποιε μονάδε, οι Γάλλοι κάποιε μονάδε. Βεβαίω υπάρχουν λοιπόν ταξίες. Πρέπει να το αντιμετωπίσουμε όπω και στη Σομαλία, Θέτοντα κάποιε προποθέσει. Δεν αρκεί να εκπαιδεύει του στρατιώτε, πρέπει να του πληρώνει κιόλα. Αλλιώ θα φύγουν. Στη Σομαλία το αντιμετωπίσαμε. Πρέπει να υπάρχει δομή διοίκηση και ελέγχου. Βεβαίω, στη Σομαλία το επιτύχαμε μέσω των Αφρικανικών δυνάμεων. Και εδώ λοιπόν πρέπει να αντιμετωπίσουμε αυτό το θέμα. Δεν μπορώ να σε εγγυηθώ μηδέν λιποταξίε. Αλλά πρέπει λοιπόν να αντιμετωπίσουμε όχι μόνο την εκπαίδευση αλλά και την αναδιάρθρωση, τη διοίκηση και τον έλεγχο του στρατού. Και δεν υπάρχουν ε, εύκολε απαντήσει. Δεν σα το κρύβω. Πρέπει όμως να το αντιμετωπίσουμε. Γι' αυτό θεωρώ ότι ο στρατός του Μαλή ούτως ή άλλως δεν ήταν ε, θετικό αλλά αρνητικό στοιχείο σε όλη την πολιτική διαδικασία γιατί το έλεγχαν διάφορες ομάδες που ε, αντιμάχονταν η μία την άλλη. Συνδέεται λοιπόν ε, η βελτίωση του στρατού με την βελτίωση της πολιτικής κατάστασης. Αν θέλουμε να προσεγγίσουμε τις ομάδες του Βορρά Πρέπει να έχουμε έναν ε, αξιόμαχο στρατό, γιατί άμα δεν έχει δύναμη, κανεί δεν θα σα ακούσει. Και οποιαδήποτε πύλη του προβλήματο βασικά θα είναι ένα καλό στρατό του μέλη. Πρέπει να εκπαιδεύσουμε και να αναδιαρθρώσουμε. Δεν θα είναι εύκολο, το ξαναλέω. Έχουμε, ξέρετε, όλου του στρατηγού, αλλά και νεότερους αξιωματικούς. Κάποιοι είναι ικανοί, κάποιοι συμμετείχαν στο πραξικόπημα Κάποιοι διαφωνούν με τους πραξικοπηματίες. Θα αφήσω το θέμα αυτό σε αυτούς που ξέρουν περισσότερα. Αλλά πρέπει να αντιμετωπίσουμε όλα αυτά τα θέματα. Αν όπως και στη Σομαλία καταφέρουμε να δημιουργηθούν αυτές οι ομάδες μάχη με ε, μονάδες από διάφορες περιοχές του Μαλή και όχι μόνο με στρατιώτες από τον Νότο, να βάλουμε και κάποιους του Βορρά θα δημιουργήσουμε ίσως έτσι νέες ε, δομές και μία νέα αίσθηση κοινή ε, στρατηγικής κοινού σκοπού. Πρέπει να αντιμετωπίσουμε και να χρησιμοποιήσουμε καλύτερα και τους νέους αξιωματικούς που πολλές φορές είναι πιο καλά εκπαιδευμένοι. Συνδέεται όπως είπα και με την πολιτική διαδικασία γιατί στην τελευταία ανάλυση ο λαός του Μαλή θα πάρει τις αποφάσεις. Δικός τους είναι ο βασικός ρόλος σε πολιτικό επίπεδο. Στόχος μας λοιπόν είναι να είναι ένας ικανός αποτελεσματικός στρατός που να ελέγχεται από μια δημοκρατική πολιτική κυβέρνηση. Έτσι θα αντιμετωπίσουμε το θέμα της νομιμοποίησης που θέσατε, κυρία μου. Βεβαίω έχουμε ως βάση το ψήφισμα του Συμβουλίου Ασφαλεία των ΗΠΑ που τονίζουν ότι πρέπει να γίνει αυτό, 271-285, και υπάρχει και το αίτημα των ίδιων των ε, αρχών του Μαλή να εκπαιδεύσουν το στρατό τους. Και γενικότερα ευρεία διεθνή συνένεση ότι αυτά πρέπει να γίνουν. Αλλά συνδέεται με την πολιτική διαδικασία. Οι πρόοδοι, οι επιτυχίες ε, στο πεδίο τη μάχη πρέπει να συνοδευτούν από προόδου στο πολιτικό επίπεδο. Γι' αυτό θα δημοσιεύσουμε σύντομα και θα επιχειρήσουμε να εφαρμόσουμε σύντομα τον οδικό χάρτη. Ξαναλέω, περίπλοκα θέματα, περίπλοκες απαντήσεις. Είπατε ότι εξεπλάγημεν ορισμένοι. Υπενθυμίζω ότι και στην Επιτροπή εδώ και στην ΑΦΕΤ είχαμε πει ως υπηρεσία εξωτερικής ε, ε, δράσης ότι υπάρχουν προβλήματα για τη Λιβύη και γενικότερα για την περιοχή. είχαμε πει ότι χρειαζόταν μια ε, τέτοια αποστολή στρατιωτική, γιατί μόνο στρατιωτική αποστολή μπορεί να ε, λειτουργήσει σε ένα τέτοιο τεράστιο ε, χώρο που είναι μάλιστα και έρημος. Αναφερθήκαμε επίσης σε όλες αυτές τις ροές μέσω της Γουνές βισάου. αναφερθήκαμε στο εμπορία ανθρώπων Και τα κράτη-μέλη έλεγαν μάλιστα, το γνωρίζουμε, αλλά κανείς δεν έμοιαζε, έμοιαζε να ανησυχεί τόσο πολύ. Βέβαια η κατάσταση άνοιξε στη, άλλαξε με τις εξελίξεις στη Λιβύη, όπου είδαμε ότι ε, ε, κάποιες δυνάμεις του Καντάφη πέρασαν στους Τουαρέ και αντίστροφα. Άλλαξε λοιπόν η ισορροπία δυνάμεων στην περιοχή. Έχουμε επίση αποστολή, είπα και προηγουμένω, στο Νιζέρ, που την προτείναμε και στις αρχές του Μαλή για να τους βοηθήσουμε να καταπολεμήσουν την τρομοκρατία. Αλλά κάπως χλιαρά το αντιμετώπισαν λέγοντας ε, ναι καλά γιατί όλοι ήξεραν ότι η ουσία του προβλήματος είναι το πρόβλημα των Τουαρέγ. Υπήρξε λοιπόν έγκαιρη προειδοποίηση κάποια προμηνύματα καλύτερα, αλλά μόνο όταν άλλαξε η κατάσταση στη Λιβύη άλλαξε ριζικά η κατάσταση. Βεβαίω έχουμε και άλλα σημαντικά προγράμματα. Αλλά δεν μπορούν πάντα εύκολα να εφαρμοστούν. Το ίδιο και με την αναπτυξιακή συνεργασία. Έχει λάβει σημαντικούς πόρους από την Ένωση, το Μαλί και από κράτη-μέλη. Για το Βέλγιο ήταν κύρια χώρα χορήγησης βοήθειας. Παρ' όλα αυτά τα προβλήματα δεν λύθηκαν. Και το πόρισμα για μένα είναι ότι πρέπει να υπάρχει μια ευρύτερη προσέγγιση, όχι μόνο στρατιωτική και πολιτική και διάσταση ασφάλειας. Όλα τα θέματα πρέπει να αντιμετωπίζονται εκ παραλίλου. Μακροπρόθεσμη προσπάθεια, βεβαίως, χρειάζεται, οπωσδήποτε. Και δεν θα τα κάνει όλα η Ένωση. Η Ένωση θα αναλάβει ορισμένους τομείς αλλά και οι Αφρικανικές δυνάμεις και η Αφρικανική Ένωση και το ECOWAS θα πρέπει να κάνουν πολλά. Για παράδειγμα στο Βορρά. Αλλά οι περιοχές που θα απελευθερωθούν από τις ε, γαλλικές, ε, από τις δυνάμεις του Μαλή, κατόπιν από άλλες αφρικανικές δυνάμεις, πρέπει να δούμε πώς θα εγκαταστήσουμε διακυβέρνηση, αλλά και ανάπτυξη, κάποιες αλλαγές, ούτω ώστε να διασφαλίσουμε ότι θα αλλάξει η ζωή των ανθρώπων. Πολλά πρέπει να γίνουν ε, και στον πολιτικό τομέα. Πρέπει να αλλάξει η νοοτροπία εκεί. Ελπίζω να απάντησα στα περισσότερα, ίσως όχι σε όλα, αλλά να επανέλθω κατόπιν. Ο Ναύαρχος Βουίλιαμς θα πάρει το λόγο, εν συνεχεία θα αντιδράσουν οι συνάδελφοι στα όσα είπατε. Κύριε Williams, να προσθέσω και εγώ μερικά σημεία. Σε αυτά που είπε ο κύριο Νταφ για την αποτυχία του στο επίπεδο των πληροφοριών. Ξεκινήσαμε στις ε, αρχές ε, του χρόνου ε, με την MNLA στην αντιπολίτευση και εν συνεχεία καταλήξαμε η MNLA να είναι υπόδουλη της αντιπολίτευσης. Δηλαδή, η αντιπολίτευση αποτελείται από διάφορες δυνάμεις με διαφορετικούς σκοπούς και επιδιώξεις. Τελικά τον Ιανουάριο άλλαξαν τα δεδομένα. Το να εντοπίσουμε πότε ακριβώς θα γίνει, όμως και να το προβλέψουμε ήταν πολύ δύσκολο. Εύκολο να το λέμε εκ των υστέρων. Αυτό συνδέεται και με τις λιποταξίες. Πάντα ανησυχούμε για τη δική μας κατάσταση. Αλλά μην ε, ξεχνάτε το ίδιο πρόβλημα αντιμετωπίζει και η αντιπολίτευση. Αυτή τη στιγμή ε, έχουν πρόβλημα λόγω της ε, γαλλικής επέμβασης. Αυξήθηκαν μεν οι δυνάμεις τους, αλλά οι περισσότερες δυνάμεις προήλθαν από άτομα που αναγκάστηκαν να ενταχθούν. Όταν άρχισαν όταν άρχισαν να δέχονται επιθέσεις, πολλοί από τους ανθρώπους τους λιποτάχτησαν. Ε, υπήρξαν λιποταξίες προς το MNLA. Το MNLA δήλωσε ότι είναι υπέρ των διαπραγματεύσεων. Το πρόβλημα είναι σύνθετο. Έχουν και αυτοί πολλά προβλήματα και έχουν και διαφορετικούς στόχους και φιλοδοξίες. Μέχρι στιγμής θα μπορούσαμε να πούμε ότι οι κινήσεις τους ήταν συμβατικές, παραδοσιακές. Τώρα όμως θα πρέπει να κάνουν πιο αντισυμβατικές κινήσεις για να πετύχουν τους ε, στόχους τους. Σε καμία περίπτωση δεν τα λέω αυτά έτσι με άνεση, με σιγουριά. Πάντα πρέπει να προσαρμοζόμαστε στα νέα δεδομένα. Δεν είμαστε μάντες. Για τις λιποταξίες πάντα. Από τη Σομαλία διδαχθήκαμε πώς μπορούμε να εξασφαλίσουμε την πίστη των στρατευμάτων. Μπορούμε να κάνουμε το ίδιο και στο Μαλή. Η συνολική μου εκτίμηση για το Μαλή είναι ότι παραδοσιακά ήταν πιο ανεκτική κοινωνία, πιο σταθερό κράτος και μόνο πρόσφατα ε, αντιμετώπισε προβλήματα. Αυτό τώρα παραπέμπει σε ένα άλλο ερώτημα. ότι οι Αφρικανοί δεν γνωρίζουν οι μεν τους δε. Μην ξεχνάτε ότι το ΕΚΟΒΑΣ, όπως είχε δημιουργηθεί από την αρχή, θεωρούσε ότι ο Μαλινέζικος στρατός ήταν βασικό συστατικό της, του αξιόμαχού του. Σίγουρα πρέπει να βοηθήσουμε το Μαλινέζικο στρατό και η Ευρωπαϊκή Ένωση θα θα σταθεί πίσω από την Αφρικανική Ένωση, ούτως ώστε να βοηθήσει, και το έχει κάνει και στο παρελθόν, να βοηθήσει λοιπόν την Αφρικανική Ένωση, ούτως ώστε να αναπτύξει την δυναμικό στρατιωτικό Πρόκειται για μια ολόκληρη διαδικασία. Ε, δεν είμαστε μόνο εμείς ε, πίσω από αυτή τη διαδικασία, αλλά και οι Αφρικανοί. Η Αφρική ανήκει στους Αφρικανούς, ούτως ή άλλως. Ε, περί αυτού πρόκειται. Συνοπτικά, μπορείτε να πείτε ότι υπήρχε μια αποτυχία στο επίπεδο των πληροφοριών, αλλά δεν πρέπει να υπεραπλουστεύουμε τα πράγματα. Οι λιποταξίες, πιστεύω ότι έχουμε ένα μηχανισμό ο οποίο θα δώσει καλά αποτελέσματα και σε σχέση με τους Αφρικανούς πρέπει να τους βοηθήσουμε να ξανακερδίσουν αυτά που είχαν, να τα αναπτύξουν, ούτω ώστε να δημιουργηθεί ένα, μια αποτελεσματική διακυβέρνηση για το Μαλί. Για την, τον ειδικό εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στο, Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων ε, στις 17 Ιανουαρίου η Κάθη Άστον κάλεσε τα κράτη-μέλη ε, να πούν τις απόψεις τους. Τώρα επιταχύνουμε τις προσπάθειες για να, υιοθετηθεί, να διορίσουμε αυτόν τον ειδικό εκπρόσωπο. Έχουμε ένα συντονιστή στο μεταξύ για τα στρατεύματα, στο Σαχέλ, που παίζει αυτό το ρόλο του ειδικού εκπροσώπου της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εμένα δεν με απασχολεί αυτό, λέει ο πρόεδρος Ντόνσου. Έχουμε ένα επικεφαλή τη επιχείρηση, ε, ένα συντονιστή εδώ, έχουμε, θα έχουμε κι άλλον εκπρόσωπο το πρόβλημα δεν είναι ότι λείπουν τα άτομα, το πρόβλημα είναι ότι λείπει η πολιτική βούληση. Ε, σε σχέση με αυτό που είπε ο κύριος Στίβενς, η, τα σημάδια που είχαμε, φυσικά τα είχαμε. Ξέρουμε πολύ καλά ότι κάθε τρεις μήνες μιλούσαμε για την κατάσταση του Σαχέλ. Πάνω από 20 συμβούλια γενικών υποθέσεων από την ε, υιοθέτηση της στρατηγικής του Σαχέλ ε, το 2011 μίλησαν για αυτό το θέμα. Όταν έχουμε έναν ύπατο εκπρόσωπο που έρχεται σε όλα τα Ευρωπαϊκά Συμβούλια και εξωτερικών υποθέσεων και λέει έχουμε αυτά τα θέματα, αλλά μην ξεχνάτε ότι έχουμε και μια στρατηγική για τη Σαχέλ που είναι προτεραιότητα, κάποια στιγμή θα πρέπει να δίνει και αποτελέσματα. Στην πραγματικότητα τα κράτη-μέλη δεν ξέρουν τι τους γίνεται. Αδιαφορούν πλήρως εκτός από κάποια και δεν νομίζω, ότι και στις Βρυξέλλες τα θεσμικά όργανα είχαν την πραγματική επιμονή ούτω ώστε να πιέσουν για αυτό το θέμα, να το βάλουν στην μερίσια διάταξη όταν χρειαζόταν. Τα λέω έξω τα δόντια, είμαι αυστηρός, το ξέρω. Έχω την εντύπωση ακούγοντάς σας ότι η υπηρεσία αυτή δεν είναι υπηρεσία εξωτερικής δράσης αλλά εντοπισμού των προβλημάτων, των απειλών, των προγραμμάτων, των συνομιλητών. Εντοπίζουμε τι μπορεί να γίνει και στο τέλο, στην τελική, τι γίνεται. Εντάξει, δεν αμφισβητώ ότι υπάρχει καλή θέληση και ότι υπάρχει μεγάλη αφοσίωση από πολλά άτομα του, της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Εξωτερικής Δράσης, αλλά δεν υπάρχουν αποτελέσματα. Υπάρχουν διάφοροι λόγοι, τοπικοί λόγοι, δεν μπορούμε να κάνουμε δράσεις ε, σε αυτές τις χώρες όταν τις θέλουν αυτές οι χώρες. Και υπάρχει σύγχυση όντω σε θεσμικό επίπεδο σε αυτές τις χώρες. Στη Λιβύη, στο Μαλή είναι μια περιοχή που αντιμετωπίστηκε προβλήματα. Και είναι πολύ άνηση η περιοχή αυτή. Όλα αυτά που ακούσαμε σήμερα το πρωί ήταν πολύ λογικά. Όλε αυτέ τι προσπάθειε είναι αξιέπαινε, πρέπει να τι ενθαρρύνουμε. Παρ' όλα αυτά έχουμε το αίσθημα ότι ακούμε πράγματα, τα ακούμε εδώ και χρόνια, τα ίδια και τα ίδια, αλλά δεν βλέπω πώ θα περάσουμε τι διαπιστώσει στι δράσει. Ζητώ συγγνώμη που είμαι τόσο αυστηρό, αλλά πραγματικά έχω αυτή την αίσθηση. Τσάρλ, έχει το λόγο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Συμφωνώ μαζί σας ότι είναι πρόκληση για την κάθε άστον να θέσει προτεραιότητες. Από, έχουμε την εξωτερική πολιτική, τα ανθρώπινα δικαιώματα και την ασφάλεια. Πώς θα τα παντρέψει όλα αυτά μαζί. Είναι μια πραγματική πρόκληση. Η υπηρεσία εξωτερικής δράσης ε, είναι τελικά Ευρωπαϊκή Υπηρεσία ε, Αντίδρασης για τα εξωτερικά θέματα. Τέλο πάντων, α μην του επικρίνω γι' αυτό. Γι' αυτά που είπε ο κύριο Westcott Πέστε μας λίγο περισσότερα για τη χρηματοδότηση. Είναι πολύ σημαντική η χρηματοδότηση. Αναφέρατε το οργανωμένο έγκλημα, τους ομήρους κτλ. Είμαστε στο... ακόμα στη φάση της ε, γαλλικής στρατιωτικής ε, παρέμβασης. Ε, λένε ότι οι Αρέγ έφυγαν από τη Λιβύη, πήραν όπλα, μετά τους α, κατέλαβαν ουσιαστικά οι τζιχαντίς. Ε, νομίζω ότι οι ίδιες ομάδες που σκότεσαν τον Αμερικανό ε, πρέσβη στο Μπενγκάζι που πήραν α, λεφτά από χώρες του κόλπου είναι οι ίδιες ομάδες και στη Λιβύη και στο Νότο μπαίνουν λεφτά από τον κόλπο σε σαλαφιστικές ομάδες. Υπάρχουν διάφορε φιλικέ ομάδε στην Σαουδική Αραβία και τα λοιπά που έχουν απεριόριστο χρήμα. Μπορούν να χρηματοδοτούν αυτέ τι ομάδε. Πρέπει να εξασφαλίσουμε ότι αυτέ οι σαλαφιστικέ ομάδε δεν θα παίρνουν λεφτά από, την, από τον κόλπο και τη Σαουδική Αραβία. Ο Αραβικό Σύνδεσμο, η GCC και ο OAC τι είπε για την ε, επέμβαση στο Μαλί, γιατί δεν είδα τι άποψη έχουν αυτές οι οργανώσεις ε, για την παρέμβαση. Ο Γκάλερ. Ε, Ευχαριστώ. Δεν θα ήθελα καθόλου να επικρίνω τις ευρωπαϊκές μας δομές και θετικά όργανα και δεν επικρίνω αυτό που κάνετε εσείς συγκεκριμένα θαυμάσια επιτελείτε τα καθήκοντά σας και εντοπίζετε όπως σωστά είπε ο κ. Ντανζάν που είναι το πρόβλημα, που είναι η πρόκληση και μετά σε πολιτικό επίπεδο πρέπει να ληφθούν οι αποφάσεις. Και βεβαίως, αν είναι θέματα στρατιωτικά, ε, είναι θέμα των κρατών μελών να θα συμμετάσχουν. Και πολιτικά λοιπόν έχω την υποψία ότι δυστυχώς δεν υπάρχει αρκετή διαθεσιμότητα, αρκετή ετοιμότητα. Βεβαίως έχουμε τις δομές και για τις ομάδες μάχης όπως μας είπατε, κανείς δεν ζήτησε να ε, αναπτυχθούν. Στην απόφαση του Συμβουλίου στο 2 της 17ης Ιανουαρίου με επιστολή της 18ης ε, Ενάτου 12, ο πρόεδρος της ε, κυβέρνησης του Μάλι ζήτησε την στήριξη της Ένωσης για να αποκατασταθεί η εδαφική ακαιρεότητα του Μαλί. Δεν ζήτησε συγκεκριμένα ποιε στρατιωτικές δυνάμεις θα πάνε, αλλά μπορούμε στα πλαίσια των δυνάμεών μας να τους βοηθήσουμε, να ανταποκριθούμε 18 Σεπτεμβρίου ήταν αυτή η επιστολή. Ερώτηση συγκεκριμένα. Εσείς τους είπατε, έχετε δυνατότητα να χρησιμοποιήσετε αυτή την ε, ομάδα μάχης. 1500 στρατιώτες. Πεζικό. Εφόσον οι Γάλλοι είναι στην πρώτη γραμμή και επειδή είναι τόσο μεγάλο το μήκος του μετόπου και οι αποστάσεις, θα μπορούσαν μεταξύ της πρώτης γραμμής και του Μπαμάκο να ε, εγκατασταθούν και να βοηθήσουν αυτές οι ομάδες μάχης. Στα κράτη-μέλη τους είπατε τι δυνάμεις έχετε, τους προσφέρατε αυτές τις δυνάμεις. Και αυτοί σας απάντησαν όχι, γιατί το Μαλί σίγουρα δεν είπε όχι, αφού ζήτησε. Ε, εσείς βεβαίως κάνετε τη δουλειά σας, εντοπίζετε τις προκλήσεις. Επιμένω ότι η κυρία Άστον, εάν δεν καταφέρνει να έχει ε, ανταπόκριση στην, ε, στο εσωτερικό των συναντήσεων αναμένω να μιλήσει δημοσίω και να πει αυτά πρέπει να γίνουν και τότε θα πρέπει τα κράτη-μέλη να πούνε μα δεν είναι και τόσο προτεραιότητά μας. Το πρόβλημά μου είναι ότι φέρεται να φταίει η Ευρωπαϊκή Ένωση ενώ για αυτά τα στρατιωτικά θέματα ε, φταίνε τα κράτη-μέλη κυρίως. Και γι' αυτό πρέπει σαφώς να πείτε μα τους είπαμε να τα μέσα που διαθέτουμε και αυτοί μας είπαν άσε δεν πειράζει. Ευχαριστώ. Κύριε Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι, θα έχουμε την ευκαιρία να συζητήσουμε ακόμα περισσότερο όλα τα ερωτήματα που έθεσε ο κύριος Ντενζόν όταν ετοιμάσουμε την αξιολόγηση της ε, δράσης της υπηρεσίας εξωτερικής δράσης. Δεν συμφωνώ με όλα αυτά που είπατε κύριε Ντενζόν. Δεν νομίζω όμως ότι όλα αυτά πρέπει να τα πούμε εδώ. Θα τα συζητήσουμε αργότερα. Ο συνάδελφος Γκάλερ έχει δίκιο πολύ ότι η ευθύνη των κρατών μελών είναι τεράστια. Η υπηρεσία εξωτερική δράση δεν μπορεί να κάνει τίποτα εάν τα κράτη-μέλη κολυσιεργούν και δεν κάνουν τίποτα, δεν την αφήνουν να δράσει. Ίσως δεν χρειάζεται πάντα να υπάρχει επίσημη συμφωνία, επίσημη συνένεση, αλλά τουλάχιστον χρειάζεται να μην υπάρχει επίσημη αντίρρηση. Γιατί σε αυτήν την περίπτωση είναι πολύ δύσκολο να δράσει η υπηρεσία εξωτερική δράση. Αυτό μην το ξεχνάμε. Αυτό ήταν το πρώτο. Δεύτερον, μια παρατήρηση που νομίζω έχει κάποια σημασία. Η περιοχή του Σαχέλ είναι προβληματική. Ήταν πάντα προβληματική. Η απερίμωση, ε, μεγαλώνει η έρημος, ε, αυξάνεται η φτώχεια, και σε πολλές πρωτεύουσε εδώ στην Ευρώπη ε, δεν καταλάβαμε ότι αλλάξανε τα, πράγματα. Ε, το Σαχέλ παρέμενε προβληματικό, αλλά με διαφορετικό τρόπο από ό,τι ήταν πριν από δεκαετίες. Σα φαίνεται κοινικό αυτό που λέω, αλλά παίζει ρόλο. Ναι, πάντα λέγαμε το Σαχέλ ήταν πάρα πολύ δύσκολο, προβληματική περιοχή, ό, η φρικτή άμμος κτλ. Αλλά άλλαξαν πολλά πράγματα και ξαφνικά το συνειδητοποίησαμε. Δεν έχω κανένα λόγο να αμφισβητήσω, αλίμονο, την αλήθεια των όσων ακούσαμε χθε. Ότι δηλαδή το θέμα του Μαλή μέχρι στιγμής ποτέ δεν είχε συζητηθεί σε δημόσια συνεδρίαση του ΝΑΤΟ. Συζητιέται μόνο στους διαδρόμους ή συζητιόταν μόνο στους διαδρόμους. Μας παρουσίασαν τα πράγματα με κάποιες υπερβολές, εντάξει. Αλλά τελικά νομίζω ότι δεν είχε ανησυχήσει πολύ τον κόσμο. Τουλάχιστον δημόσια. Δεν είχε προκαλέσει ανησυχίες. Και το λέω αυτό γιατί έρχεται σε αντίθεση με την κλασική μας τάση, που είναι διαφορετική. Διερωτώ λοιπόν, ε, μήπως αυτά που ακούστηκαν και που ακούστηκαν και χθε, μήπως όλα αυτά οφείλονται στο γεγονός ότι το ΝΑΤΟ και επομένως και τα κράτη-μέλη του ΝΑΤΟ ε, είπαν ότι η Αφρική, με εξαίρεση το θέμα της πειρατείας, είναι πρόβλημα της Ευρώπης και όχι για πρόβλημα των υπολείπων μας. Και αν αυτό είναι αλήθεια, θα πρέπει να δούμε ποιε είναι οι συνέπειε που είναι σοβαρές. Δεν είναι θέμα πολιτικών προτεραιοτήτων μόνο, έτσι, και τότε πρέπει να ανοίξουμε τα χαρτιά. Εγώ είμαι από αυτούς που εδώ και χρόνια λένε ότι υπάρχει ένας ανταγωνισμός μεταξύ του ΝΑΤΟ και αυτή την ευρυονική ευρωπαϊκή πολιτική άμυνας. για τις ομάδες μάχης. Μέχρι στιγμής δεν χρησιμοποίησαμε αυτές τις ομάδες μάχης, πιστεύω, γιατί δεν μπορούμε να τις εντάξουμε στο διοικητικό μηχανισμό του στρατού. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό. Δεν ξέρουμε πού θα τις εντάξουμε διοικητικά, δηλαδή, πού ανήκουν. Στη στρατιωτική ιεραρχία. Διστάζουμε να χρησιμοποιήσουμε μια ομάδα όταν δεν ξέρουμε πού εντάσσεται ακριβώς. Πώς διοικείται. Είναι σωστό αυτό. Είναι λάθος. Εξηγεί πάντως γιατί οι ομάδες ε, μάχης παραμένουν εκτός. Ε, τις έχουμε στη διάθεσή μας, αλλά δεν τις εντάσσουμε. Σαν το Eurocore, που είναι επίσης ένα μεγάλο κομμάτι αλλά ποτέ δεν το χρησιμοποιούμε. Α, αν δεν τα χρειαζόμαστε αυτά τα, αυτές τις ομάδες, ας τα βάλουμε στο μουσείο. Αλλά το να τις έχουμε μόνο για να τις χαιρετούμε, ας πούμε, δύο φορές ε, το χρόνο ή δύο φορές ανά κοινοβουλευτική θητεία, δεν έχουν κανένα... Δεν έχουν κανένα νόημα. Ε, το Eurocore εμείς δεν το χρησιμοποιήσαμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά το χρησιμοποίησε το ΝΑΤΟ. Και αυτό είναι το παράδοξο. Η Φρανσίσκα. Σας ευχαριστώ. Εγώ θα ήθελα να ξεκινήσω για τις λιποταξίες στη γερμανική περίπτωση. Είναι ένα καλό παράδειγμα, γιατί όπως ξέρετε ο γερμανικός στρατός έχει αλλάξει από υποχρεωτική θητεία, έχει εθελοντέ εθελοντές μόνο και το ποσοστό λιποταξίας είναι 33% μέσα στο πρώτο έτος και τώρα το ξανασκέφτονται ε, για παράδειγμα να μην ε, κάνουν πια την ε, εποπτεία με τον ίδιο τρόπο, τους εξοπλισμούς κτλ. Είναι πολύ ενδιαφέρον και γίνεται προσπάθεια να χαμηλώσει το ποσοστό λιποταξίας το οποίο είναι πολύ ψηλό αυτή τη φάση. Ο κύριο Τάνοκ εκτό μικροφώνου. Είναι ενδιαφέρον λοιπόν να δούμε το πώς κανείς ε, πρέπει να ξανασκεφτεί το θέμα της στρατιωτικής θητείας. Οι Γερμανοί έχουν επίση εκπαιδεύσει τον Μαλινέζικο στρατό. Δεν είναι μόνο οι Αμερικανοί και το πρόβλημα ήταν όντω ελέγχου και διοικησή και περισσότερο παρά δυνατοτήτων. Ιδιαίτερα οι νεότεροι φαίνεται ότι είναι καλά εκπαιδευμένοι, αλλά η διοίκηση και ο ελεγχό του είναι προβληματικό. Και με ανησύχησε κάπως το ότι είπατε ότι δεν το γνωρίζουμε ακόμα ποιο θα είναι επικεφαλής. Ε, είναι ανησυχητικό να μην έχετε ακόμα απάντηση σε αυτό. Δεύτερη παρατήρηση που ήθελα να κάνω είναι ότι φυσικά πολλοί από τους σπόρους της χώρας δεν ωφελούν τον πληθυσμό της, ανεξάρτητα από την εθνότητα κτλ. Και θα ήθελα επίσης να τονίσω ότι αυτή τη στιγμή το Κοινοβούλιο και τα κράτη-μέλη διαπραγματεύονται για τον νόμο περί διαφάνειας. Το είχαμε εδώ και στο Κοινοβούλιο όσον αφορά τους κανόνες διαφάνειας για τις δικές μας εταιρείε που έχουν έδρα στο εξωτερικό. Και υπάρχει μια κίνηση από πλευρά των μελών να αποδυναμωθούν οι απαιτήσει προς τις εταιρείε. Και το Μαλί είναι ένα υπέροχο παράδειγμα για τον ε, μπορέσουμε να πάρουμε περισσότερες ευθύνες, να αναλάβουμε περισσότερε ευθύνε από πλευρά μα. Ίσως θα έπρεπε λοιπόν να είναι ένα θέμα και αυτό. Κάτι ακόμα που θα ήθελα να σας ρωτήσω είναι ε, τα λίτρα και οι όμοιροι. Το 2003 η Γερμανία πλήρωσε τα πρώτα ε, λίτρα υπό την τότε κυβέρνηση την οποία γνωρίζω καλύτερα και πιστεύω πως ήταν ένα τεράστιο λάθος που αρχίσαμε να δίνουμε χρήματα αλλά υπήρξε πολιτική όλων των ευρωπαϊκών κυβερνήσεων στην περιφέρεια αυτή να ε, πληρώνουν τα λίτρα. Και αυτό πιστεύαμε υπάρχει αλλαγή στην ευρωπαϊκή πολιτική που να λέει ότι δεν το χρειαζόμαστε πλέον γιατί στην ουσία αγοράζουν όπλα και με αυτά τα χρήματα δεν βοηθά σε τίποτα και όπως βλέπουμε δέκα χρόνια μετά δεν είναι καθόλου καλή η πολιτική. Μήπως θα έπρεπε μαζί όλοι να αλλάξουμε πολιτική. Υπάρχει σχετική συζήτηση ανάμεσα στα κράτη-μέλη και έπειτα για τα όσα είπε ο κύριος ε, ε, ε, Τάνοκ για τα χρήματα της Σαουδικής Αραβίας και του Κατάρ που πάνε εκεί. Η ε, Γερμανία εξάγει ε, πάνζερ στην Σαουδική Αραβία. Μα δεν θα πρέπει να το κάνουμε εφόσον χρηματοδοτούν αυτού του ανθρώπου που στην ουσία υπονομεύουν του δικού μα στόχου στην περιοχή. Θα πρέπει να τα συνδέσουμε αυτά και να σκληρύνουμε τη στάση μα απέναντι στη Σαουδική Αραβία και το Κατάρ και να μην παριστάνουμε ότι δεν συνδέονται αυτά τα θέματα μεταξύ του. Και θέλω να αντιδράσω σε ένα από τα ερώματα που έδειξε ο κύριος Ντανζάν. Το φθινόπωρο του 2012 η κυρία Γκισάρ εστάλει από την Ευρωπαϊκή Ένωση για να εντοπίσει τι μπορούμε να κάνουμε στο Μαλί. Υπήρχε ήδη δηλαδή ε, ε, μια αποστολή εντοπισμού και αξιολόγησης. Γιατί τώρα πρέπει να στείλετε νέα αποστολή. Υπήρξε μια διαδικασία τέτοια το, την Άνοιξη. Δεν γίναν όλα όπω είπατε ξαφνικά ε, και δεν ήταν κεραυνό. Τώρα πρέπει να στείλετε κι άλλη αποστολή. Τι έγινε με τα αποτελέσματα εκείνη τη αποστολή και τα πορίσματά της. Και έχω δύο ακόμη ερωτήσεις. Υπάρχουν φήμες, τουλάχιστον κυκλοφορούν στο γερμανικό τύπο, ότι η ECOWAS ζητά τη χρηματοδότηση για την ε, Αφρικανική Διευκόλυνση για την Ειρήνη και ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση το αρνείται αυτό. Είναι τελείως λάθος ή αληθεύει ότι δηλαδή η Ένωση αρνείται να χρηματοδοτήσει την ΕΚΟΒΑΣ για να παρέμβει στο Μαλί. Και η τελευταία μου ερώτηση, νομίζω πως είχατε δίκιο κύριε Στίβενς λέγοντας ότι πρέπει να δώσουμε διακυβέρνηση στις ε, περιοχές που ανακατακτώνται. Αλλά ποιο θα κυβερνήσει. Μπορείς να πας στο στάτου κουβό που, που ισχύει πριν και να πει ότι θα είναι τον Παμακό. Δεν νομίζω πως θα γίνει δεκτό. Κράτο δικαίου και όλα αυτά, ωραία λόγια. Αλλά και πάλι ποιο θα τα αναλάβει όλα αυτά. Και ε, τα όσα συμβαίνουν αυτή τη στιγμή στο Μαλί επηρεάζουν ε, τις αποστολές μας στη Λιβύη. Ευχαριστώ, Άντρου Νταφ. Μια γρήγορη ερώτηση, ελπίζω. για την Τουρκία που όπως ξέρετε συχνά ζητά συνεργασία για τον αγώνα κατά των τρομοκρατών του ΠΚΚ. Ξέρουμε ότι το ΝΑΤΟ ε, στην ουσία έχει παραλύσει πολιτικά τουλάχιστον λόγω του τουρκοκυπριακού προβλήματος αλλά θα με ενδιέφερε να ακούσω αντιδράσεις που ίσως να ακούσατε, να είχατε από την Άγκυρα. για άσκηση πολιτικής πίεσης. άσκηση πολιτικής πίεσης στους Άραβες ώστε να ασχοληθούν με το επιδενούμενο πρόβλημα του φανατισμού της τζιχάντ στο Σαχέλ. Ε, έχετε μιλήσει με τον κύριο Ταβούτογλουσε για αυτό το θέμα και για τα σχετικά προβλήματα. Euh, Μάλιστα. Θα κάνουμε ένα τελευταίο γύρο απαντήσεων. Ευχαριστώ. Να σχολιάσω για το σημαντικό θέμα που ε, το ερώτημα εκείνο που είπε αν είμαστε υπηρεσία εξωτερικής δράσης ή αντίδρασης. Εγώ ε, ε, είμαι σε αυτή την υπηρεσία εξ αρχής και εντόνως θα επιμείνω ότι είμαστε υπηρεσία δράσης. Και θέλω να υποστηρίξω για την ε, ε, είπατε εκπρόσωπο όπου για όλα αυτά τα θέματα θέλει και είναι υπέρ της διατήρησης όλων αυτών των ε, υποθέσεων στην Αφρική, που έχουμε πολλές υποθέσεις στην Αφρική και πρέπει να το διαχειριστούμε. Και από τα κράτη-μέλη, να σας πω ότι υπήρξε επιστολή από 5 με 8, 5-8 υπουργού εξωτερικών το 2010 που ζητούσαν τότε από την ύπατη εκπρόσωπο να συγκροτήσει στρατηγική για το Σαχέλ. Ήδη υπήρχε, αλλά ήταν ένα από τα πρώτα καθήκοντα που χρειάστηκε να αναλάβω, να συγκροτήσουμε τέτοια στρατηγική, να την θέσουμε επιτάπητος και να την υποβάλλουμε στα κρατημέλη που γνωρίζουν ότι είναι ε, μια ευάλωτη περιοχή. Υπάρχει το γεγονός ότι δεν συζητείται σε κάθε συνεδρίαση του, Υπουργείου του Συμβουλίου Υπουργών Εξωτερικών δεν σημαίνει ότι δεν ασχολούμαστε με το θέμα Σαχέλ. Συμφωνώ, αλλά δεν υπάρχουν πολλές κρίσεις όπου, τα όπου κάποιο κράτος μέλος έχει μπει σε πόλεμο. Ακόμα και στη Συρία δεν υπάρχει κανείς. Ευρωπαίος. Τώρα, το Μαλί προέκυψε από το γεγονός ότι έχουμε ένα κράτος το οποίο πολεμά εκεί, έχει στρατό εκεί και γι' αυτό και έγινε και έκτακτο Συμβούλιο Υπουργών Εξωτερικών αμέσως μόλις αυτό έγινε. Δεν είναι το θέμα μας σήμερα, αλλά εμείς στην Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης ήδη προετοιμάζουμε στρατηγικές σκέψεις για το πώς θα χειριστούμε την, ε, την ασφάλεια, το, την θαλάσσια στον κόλπο της Γουινέας. Είναι πρόβλημα αυτό και θα είναι και μεγαλύτερο μεγαλύτερο πρόβλημα από τη στιγμή που δεν θα το χειριστούμε, δεν θα το αντιμετωπίσουμε. Και θα σας ε, ενημερώσουμε για το τι, τι θα κάνουμε εκεί και τα όσα συμβαίνουν στην περιοχή των Μεγάλων Λιμνών. Ε, είναι ένα πρόβλημα που νομίζαμε ότι έχει κάπως ε, αυληθεί αλλά η κατάσταση επιδεινώνεται. Υπάρχουν δηλαδή πολλά τα οποία δεν τα βλέπετε άμεσα, αλλά για τα οποία προετοιμαζόμαστε για την ε, αλκαϊδα και τα παρακλάδια της στο Μαγρέμπ που είναι δραστήρια και ενεργή. Τι συνέβη λοιπόν εκεί ε, τώρα τον Ιανουάριο. Εντοπίσαμε πολύ γρήγορα σε πρώιμο στάδιο τη σημασία της επανεκπαίδευσης του Μαλινέζικου στρατού και τη στήριξή του με την Ευρωπαϊκή Ένωση, γιατί πιστεύαμε ότι θα ήταν πολύ σημαντικό για να μπορέσουμε να περιορίσουμε αλλά και να αναχαιτήσουμε ενδεχομένω τον ε, έλεγχο των ανταρτών στο βορρά. Πήρε πολύ χρόνο να πείσουμε τους ε, ε, Μαλινέζους και την περιοχή ολόκληρη ότι αυτό ήταν απαραίτητο. Η ECOWAS, για να είμαστε δίκαιοι, είπε ότι θέλουμε να μπούμε και να βοηθήσουμε. Όμω ε, οι Μαλινέζοι είπαν δεν χρειαζόμαστε βοήθεια από κανέναν. Εμεί θα ανακτήσουμε το βορρά μα. Αφήστε το σε εμά. Αλλά κάναν λάθο και τώρα το δέχτηκαν ότι έκαναν λάθο και ζητούν ε, ευχαρίστω τη βοήθειά μα και τη δέχονται. Ε, Κάποιε φορέ αυτά τα πράγματα παίρνουν χρόνο και γι' αυτό. Η ECOWAS βρήκε ότι και εκείνη πήρε πολύ χρόνο για να συγκεντρώσει δυνάμεις λοιπά. Και αυτοί τώρα επιτάχυναν τις διαδικασίες. Γι' αυτό και προσπαθούμε να βοηθήσουμε να χρηματοδοτήσουμε την αφίσμα. Ήδη έχουμε εντοπίσει 50 εκατομμύρια ευρώ που θα πάνε εκεί. Ε, έχουμε λάβει επιστολή του Πρόεδρου της ECOWAS πριν από 6 μήνες πάνω κάτω που έλεγε παρακαλούμε, 500 εκατομμύρια μας λείπουν για να πληρώσουμε για την αφίσμα και για να εκπαιδεύσουμε τον Μαλινέζικο στρατό. Φυσικά δεν απαντήσαμε. Αμέσως είπαμε ναι, τι τα θέλετε, δώσε μας λεπτομέρειες, δώστε μας ε, το προπολογισμό σας. Έχουμε και εμείς ευθύνε και είμαστε υπόλογοι αφού δίνουμε τα λεφτά των φορολογουμένων. Πρέπει κάπου να πούμε ότι πάνε, δεν μπορούμε να λέμε ότι τα στείλαμε στον τάδε. Λοιπόν, επανέλθετε, τους είπαμε και πείτε μας τι θέλετε να κάνετε και εμείς βοηθάμε την EcoWest να φτιάξει τις εκτιμήσεις της και τον προπολογισμό. Και όλα αυτά θα συζητηθούν ε, στην ε, διάσκεψη των δωρητών που είναι προγραμματισμένη για τις 29 στην Αντισαμπέμπα. Δεν τα χρηματοδοτήσουμε όλα εμείς. Οι ήδη είπαν ότι κάποια χρήματα θα δώσουν. Ίσως και κάποιες χώρες του Περσικού κόλπου να είναι έτοιμες να συμβάλλουν επίσης. Ε, τώρα εδώ υπάρχει και ένα ενδιαφέρον ερώτημα Λοιπόν, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα, η Τουρκία, η Αίγυπτος έχουν θίξει κάποια ερωτήματα. Καταρχήν, όλα τα μέσα της διεθνούς κοινότητας, το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ, όπως και η Ένωση, έχουν ενεργήσει ομόφωνα για όλα αυτά και οι εκπρόσωποι της Μέσης Ανατολής, οι περιφερειακοί εκπρόσωποι στο Συμβούλιο Ασφαλείας, ομόφωνα η Ρωσία, η Κίνα στήριξαν αυτή την επέμβαση. Γιατί ανταποκρίνεται σε ένα θεμητό νόμιμο αίτημα των νομίμων αρχών που αντιπροσωπεύουν το λαό του Μαλή. Ε, εμείς είμαστε εκεί λοιπόν, η Ένωση είναι εκεί για να στηρίξει το λαό του Μαλή. Όποιος ε, το επικρίνει αυτό, αναρωτιέται κανείς με ποιανού το μέρος είναι. Μετά από τη συνεδρίαση λοιπόν που σκοπεύουμε να κάνουμε στις 5 Φεβρουαρίου που θα έχουμε εκπροσώπους της ΟΑΣΕΑ από το Συμβούλιο Συνεργασίας του Περσικού κτλ. Θα κάνουμε λοιπόν συζήτηση για το τι θέλουμε να επιτύχουμε και πώς θα το επιτύχουμε αυτό. Κανένας δεν θέλει να αμφισβητήσει τα δικαιώματα οποιοδήποτε για το Βορρά εκτός από τις τρομοκρατικές ομάδες που είναι εξαιρετικά ευχαριστημένοι να καταπατούν τα δικαιώματα όσων διαφωνούν μαζί τους. Εμείς θέλουμε, στόχος μας είναι να αφήσουμε τον λαό του Μαλή να ανακατακτήσει αυτή τη γη. Ο περσικό κόλπο και οι αραβικέ χώρε θα πρέπει να είναι παρούσει και θα συζητήσουμε μαζί του. Δεν θέλω να προκαταβάλω τα αποτελέσματα αυτού, ε, ε, αυτής Τώρα, η Αλγερία και τα λίτρα. Οι Αλγερινοί δεν πληρώνουν λίτρα. Έχουν τέτοια πολιτική όπως γνωρίζετε και είδατε. Κάθε χώρα τώρα έχει μια ευθύνη απέναντι στους πολίτες της. Να Έχει καθήκον να προστατεύει, να προστατεύει τη ζωή τους στο εξωτερικό. Αλλά κατά πόσο τώρα τα... η πληρωμή λίτρων στην ουσία ωφελεί τους απαγωγείς, αυτό είναι θέμα κάθε κράτους μέλους. Ευχαριστώ. Yes, also Ένωση, δράση, αντίδραση κτλ. Ποιος καθορίζει τα προβλήματα. Πολλά γίνονται που τα κάνει κάθε άστον και που δεν τα γνωρίζει η κοινή γνώμη. Αλλά κοιτάξτε, το θέμα αυτό είναι η ιδιοκτησία των Αφρικανών. Και έχουμε συζητήσει με εκπροσώπους του Μαλή για τη στρατηγική μας και ο πρέσβης του Μαλή όταν το συζητήσαμε κάποια φορά μαζί του μας είπε βεβαίως, βεβαίως ευχαριστούμε αλλά πρέπει να συνεργαστείτε μαζί μας και εμείς θα παίξουμε τον ηγετικό ρόλο. Οι χώρες αυτές, ε, Αλγερία, Νιζέρ, Μάλι, ε, συζητούν μεταξύ τους και προσπαθούν να καταλήξουν Αυτές ε, είναι χώρες που, τις οποίες δεν μπορούμε να πιέσουμε. Προτείναμε κάποιες άλλες το στο Μαλί και μας είπαν ναι θα το δούμε αλλά ποτέ δεν μας είπαν ε, οριστικά ναι. Είναι κυρίαρχα κράτη πρέπει να το λάβουμε υπόψη. Είναι περίπλοκα τα θέματα. Δεν μπορείτε να δώσετε απλοϊκές απαντήσεις δεν μπορούμε να στείλουμε τις δυνάμεις μας ε, να πάνε στην α ή τη β περιοχή. Δεν θα το εκτιμήσουν οι Αφρικανοί οι ίδιοι. Όχι λοιπόν απλοϊκές απαντήσεις. Πολλά έγιναν. Για πρώτη φορά στις 19 Οκτωβρίου το ΕΚΟΒΑΣ και η Αφρικανική Ένωση που προηγουμένως ε, ήταν ε, ο ένας κατά του άλλου η Ευρωπαϊκή Ένωση ή τα Ενωμένα Έθνη Όλοι πήγαν στον Παμακό και είπαν πρέπει να γίνει αυτό ο δικός χάρτης, να προσεγγίσουμε τον Νότο, να βελτιώσουμε τον ε, στρατό του Μαλή και την ε, διακυβέρνηση. Και η Ένωση το υποστηρίζει. Και όχι απλώς το υποστηρίζει, αλλά δρά έγινα συνεδριάσει εδώ στις Βρυξέλλες με εκπροσώπους των Εθνών, με τον κύριο Πρόντι, για να υλοποιηθεί η στρατηγική μας. <clears throat> δεν τα βλέπετε σωστά αυτά, δεν τα γράφουν εφημερίδες, δεν είναι τόσο ε, γαργαλιστικά θέματα, αλλά <clears throat> βεβαίως και εγώ έναντι της κυβέρνησής μου μπορώ να πω <clears throat> γιατί δεν στείλατε στρατό να πολεμήσει τους ε, τρομοκράτες. Αλλά είναι, επαναλαμβάνω, κυρίαρχα κράτη, είναι αφρικανικά θέματα αυτά για τις ομάδες μάχης. Ε, δεν θέλω να καλυφθώ λέγοντας δεν Μα υπευλήθη έτοιμα. Όντω δεν μας υπευλήθη έτοιμα. Αλλά εμείς είχαμε κάνει τον προγραμματισμό. Αλλά βεβαίως ε, πρέπει να ελέγχεις πάντα και τις διάφορες μονάδες τη ομάδα μάχης. Και ναι, μεν δεν έχει τεθεί επισήμω ε, στην ημερήσια διάταξη, αλλά έχουν γίνει διαβουλεύσει. Πρέπει να υπάρχει πολιτική βούληση των χωρών που ε, έχουν τις ε, μονάδες που συγκροτούν την ομάδα μάχης. Κάποιες ήταν πιο έτοιμο πόλεμες, κάποιες όχι. Αλλά δεν έχει τελειώσει η συζήτηση για το θέμα αυτό. Θα υπάρξει και μια φάση σταθεροποίηση όπου θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν οι ομάδες μάχης. Ευρύτερα βεβαίως και εν ώψη του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου θα το ξαναδούμε αυτό το θέμα των ομάδων μάχης. Το ερώτημα είναι είναι ε, για επιχειρήσεις ή είναι μόνο για να διαμορφώνει την κατάσταση και για να ε, μεταδίδεται η γνώση. Θα το εξετάσουν λοιπόν οι Υπουργοί. Οπωσδήποτε και εδώ μπορούμε να το συζητήσουμε. Δίκηση και έλεγχος είναι επίσης δυσχερές θέμα. Το είπα και στην εισαγωγή μου. Είναι κινούμενος στόχος, ξέρετε είναι πολύ δύσκολο και στην ακτή του ελεφαντοστού και εκεί προσπαθούμε να αναδιαρθρώσουμε τις δυνάμεις ασφαλείας. Πρέπει να δούμε πώς θα αντιμετωπίσουμε τους υπάρχοντες αξιωματικούς ε, κάθε βαθμού, στρατηγούς κτλ. Είναι ιδιαίτερο πολιτικό θέμα. Όταν γίνονται διορισμοί ε, στρατηγών, ακόμη και στη Γαλλία και τη Γερμανία, είναι πολιτικό θέμα. Ξέρετε πολύ καλά ότι η δομή του στρατού στο Μαλί ε, αντανακλά την πληθυσμιακή σύνθεση της χώρας. Υπάρχουν, για παράδειγμα, τάγματα του ΑΡΕΓ. Θα τα κρατήσουμε έτσι, αμυγός του ΑΡΕΓ ορισμένοι από τους αξιωματικούς ε, συμμετείχαν στο πραξικόπημα. Άλλοι όχι. Όλους αυτούς πρέπει να τους συνδυάσουμε. Κινούμενος στόχος λοιπόν και ε, συνδέεται πολύ με την λήψη πολιτικών αποφάσεων. Το συζητάμε και με τους επικεφαλείς των αποστολών έχει συγκεκριμένους στόχου, έχει μιλήσει με τις πολιτικές αρχές. Πρέπει να τον παρακολουθήσουμε εκ του σύνεγγυ. Για την Τουρκία, σημειώνω, και για την Αίγυπτο εξάλλου. Καλούμε και αυτές τις ε, χώρες να συμμετάσχουν. Θα τους κάνουμε λοιπόν και στην Αίγυπτο και στην Τουρκία πρόσκληση, θα τους αποστείλουμε πρόσκληση παρά αυτά που είπαν οι πρόεδροι τους. Και ξέρω ότι κάποια από την ε, υπηρεσία εξωτερικής δράσης έχουν πάει στο Κάιρο, μίλησαν με τον Υπουργό Εξωτερικών και τους βοηθούς του Προέδρου και παρά τις δηλώσεις του Προέδρου οι Αιγύπτιοι ενδιαφέρονται, δεν ξέρω αν θα συμμετάσχουν, αλλά δείχνουν πολύ ενδιαφέρον ε, για να δουν τι θα μπορούσαν να κάνουν. Κάτι έχει γίνει λοιπόν γι' αυτό. Βεβαίως η Λιβύη συνδέεται πάρα πολύ και με τις εξελίξεις στη Συρία. Όπως ξέρετε, όπλα και δυνάμεις πήγαν από τη Λιβύη στο Σαχέλ και τώρα φοβούνται ότι θα επανέλθουν. Ανησυχούν λοιπόν πολύ για τα σύνορά τους. Σχεδιάζουμε και τα κράτη-μέλη συμφώνησαν, όχι ακόμη σε επίπεδο υπουργών, αλλά σε χαμηλότερο επίπεδο, ότι θα υπάρξει μία αποστολή για την ασφάλεια των σύνορων. Αλλά και η Λιβύη είναι κυριαρχό κράτος, ε, πολύ ευαίσθητα θέματα αυτά. Μόνο ό,τι θέλουν μπορούμε να κάνουμε δεν θέλουν να στείλουμε ολόκληρο τάγμα στα νότια σύνορά τους. Γιατί θέλουν να τα ελέγχουν οι ίδιοι. Και επιμένουν στην προστασία της κυριαρχίας τους. Και παρά το ότι η Λιβύη δεν είχε κυβέρνηση ή μετά δεν είχε κυβέρνηση και μετά είχε λίγο πάλι κυβέρνηση μέχρι τα μέσα Νοεμβρίου. Συζητήσαμε τις πολιτικές αρχές και αποδέχθηκαν την αποστολή ασφάλειας όπου θα εκπαιδεύσουμε το στρατό και τα σώματα ασφαλείας ούτως ώστε να έχουν σωστή φύλαξη των συνόρων τους και των ε, βορείων ε, θαλασσίων συνόρων και των ε, νοτίων συνόρων όπου δεν έχουμε μπορέσει να πάμε ακόμη για λόγους ασφαλείας. Όλα αυτά είναι σε φάση διαμόρφωσης. Αλλά προγραμματίζουμε λοιπόν αυτή την αποστολή. Θα είναι στην ημέρα σε διάταξη τον Υπουργών Εξωτερικών στην 31 πρώτου. Τα κράτη-μέλη λοιπόν, θέλουν να, γίνουν, θέλουν να γίνουν γρήγορα τα πράγματα, δεν θα λύσουμε φυσικά όλα τα προβλήματα. Και εδώ ψάχνουμε συνεργασίες με τη Frontex για παράδειγμα. Θέλουμε να το συνδυάσουμε με πρωτοβουλίες Frontex και άλλες πρωτοβουλίες της Κομισιόν. Είναι στα πλαίσια της ευρύτερη αντιμετώπισης μας της Λιβύης. Γιατί υπάρχει σαφώς σύνδεση. Σύνδεση ΝΑΤΟ-Ένωσης. Βεβαίως, πάντα υπάρχει κάποιος ανταγωνισμός. Αν και νομίζω ότι η θεολογική, ιδεολογική συζήτηση, ας την αποκαλέσω έτσι, έχει παρέλθει. Γίνονται συζητήσεις. Αλλά έχουν και οι δύο καταλάβει ότι μπορούμε να ε, αλληλοσυμπληρώσουμε τις, ε, τα καθήκοντά μας. Δεν λέω ότι δεν υπάρχει καθόλου ανταγωνισμός πλέον, αλλά το προσωπικό των δύο οργανισμών ε, συζητάει. Συζητάμε για το κοσφοπέδιο, της Ομαλία πώς μπορούμε να συνεργαστούμε, γιατί σε αυτές ε, τις περιοχές και σε άλλες είμαστε και οι δύο παρόντες. Αλλά αλλάζει πολύ και το στρατηγικό πλαίσιο. Η αμερικανική ε, στρατηγική ασφαλείας είπε εμείς ε, στραφόμεθα προς ε, Ανατολάς. Δεν μπορούμε να κάνουμε όλα όσα κάναμε μέχρι τώρα στην Ευρώπη. Πρέπει να αναλάβετε ένα μεγαλύτερο τμήμα των ε, καθηκόντων ασφαλείας. Αυτό θα επηρεάσει και το δυναμικό μας και το χρόνο που θα χρειαζόμαστε για να παρεμβαίνουμε. Γι' αυτό το βάλαμε στην ημερήσια διάταξη. Ο πρόεδρος Φαν Ρόμπαϊ το έθεσε στην ημερήσια διάταξη του Συμβουλίου Κορυφής Υπάρχει η βέλτιστη κατανομή ε, καθηκόντων. Δεν θα το έλεγα, αλλά το ΝΑΤΟ έχει ως κύριο καθήκον το Αφγανιστάν και στη θάλασσα γύρω από τη Σομαλία με την αποστολή ε, ασπίδα του ωκεανού που έχει πλέον μόνο ένα πλοίο και επίσης το κοσφοπέδιο. Αλλά αλλάζει και από πλευράς ε, δυνατοτήτων η κατάσταση στο ΝΑΤΟ γιατί ε, οι αμυντικέ δαπάνε είναι πολύ σημαντικέ για την Ένωση και για το ΝΑΤΟ, αλλά και η Ένωση και το ΝΑΤΟ πρέπει να προσαρμοστούν στο νέο πλαίσιο. Είναι ευρύτερο θέμα να μην πειράσω λεπτομέρειε γιατί περνάει και η ώρα. Βεβαίω πολύ σύντομα. Για το ΝΑΤΟ, λέει τώρα ο υπονάβαρχος σε επίπεδο προσωπικού έχουμε πολύ στενή σχέση με τους συναδέλφους μας στην άλλη πλευρά των Βρυξελών, όχι περιστασιακά. Καθημερινή, ωριαία συνεργασία έχουμε, όπως απαιτείται και όπως επιθυμούν τα κράτη-μέλη, για να διασφαλίσουμε ότι δεν υπάρχει ανταγωνισμός, αλλά επικοδομητικός διάλογος που προωθεί λύσεις και δεν δημιουργεί δυσχέρειες. Άλλο σχόλιο για τις ε, γερμανικές λιποταξίες. Είναι το θέμα... Μιλάγατε για καψόνια όπου δεν τους αφήνουν να κοιμηθούν κτλ. Πρέπει αυτό να γίνεται παντού, σε οποιαδήποτε εκπαίδευση. Θα το κάνουμε και όταν θα εκπαιδεύσουμε το στρατό του Μαλή. Στόχος είναι να ανταποκριθείς για να αντιμετωπίσει του αντιπάλου. Εάν δεν είσαι όσο καλό και εκείνη θα αποτύχει. Άρα εκπαιδεύει με βάση τις συνθήκε μάχη. Άρα το πόσο σκληρή θα είναι η εκπαίδευση πρέπει να προσαρμόζεται στι ανάγκε σου. Και αυτό σημαίνει ότι κάποιες φορέ πρέπει να υπερβεί αυτά που είναι συνηθισμένα στην κοινωνία. Μπορεί κάποιε προποθέσει του συγκεκριμένου στρατιώτε να είναι σκληρέ κατά την εκπαίδευση. Είμαι σίγουρο ότι επικεφαλή της ε, ομάδας εκπαίδευσης, της αποστολής εκπαίδευσης στο Μαλί ξέρει το επίπεδο εκπαίδευση στο οποίο πρέπει να υποβληθούν οι στρατιώτε του Μαλί για να ανταποκριθούν στην αποστολή του. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ. Κύριε. Είναι μια συζήτηση που δεν θα τελειώσει εδώ. Ίσως θα πρέπει να συναντιόμαστε πιο τακτικά, γιατί η κατάσταση είναι τέτοια που δικαιολογεί πιο συχνές επαφές. Υπάρχουν πάρα πολλά δεδομένα, πάρα πολλά στοιχεία έχουμε επιτάπητος. Πρέπει να ξεχερσώσουμε λίγο το έδαφος, να βγάλουμε τα άχρηστα στοιχεία, να κρατήσουμε αυτά που μας χρειάζονται. Κράτησα τα επιχειρηματά σας, τα οποία είναι βάσιμα, ότι είναι κυρίαρχα αυτά τα κράτη. Δεν μπορούμε να κάνουμε εμείς ό,τι θέλουμε, με το ρυθμό που θέλουμε στην Αφρική. Απόλυτα κατανοητό και συμφωνώ. Πολλά γίνονται με διακριτικότητα επίση, όχι φανερά, ίσως δεν τα ξέρουμε και δεν τα μαθαίνουμε αμέσω. Παρ' όλα αυτά, για αυτό το θέμα που είναι μακρόπνο, έχουμε την αίσθηση ότι πρέπει να υπάρξει μεγαλύτερη εστίαση, μεγαλύτερη δράση και αποφασιστικότητα και αυτό ξεπερνάει το πλαίσιο δυνατοτήτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και είναι και δουλειά των κρατών μελών να παίξουν το ρόλο τους και είπα ότι εκπρόσωπος είναι συνυπεύθυνοι κι αυτοί Και ό,τι δώσει. Ελπίζω να δώσει καλά αποτελέσματα. Και την επόμενη φορά που θα συναντηθούμε, κάποια από τα πράγματα που υπόθηκαν στα συμπεράσματα του Συμβουλίου, ελπίζω να μπορούν να έχουν υλοποιηθεί. Θα ακούσουμε και τον ε, στρατηγό Λεκουάντχα και ελπίζω η επόμενη φάση να προχωρήσει απρόσκοπτα. Ευχαριστώ και καλό κουράγιο. Και θα πάμε στο επόμενο σημείο της ημερήσιας διάταξης, αφού κάνουμε πρώτα ένα διάλειμμα 10 λεπτών. Euh, Αγαπητοί συνάδελφοι, Πάμε στο τελευταίο σημείο στη μέση διάταξη. Εξαγωγές όπλων. Εφαρμογή της κοινή θέσης του Συμβουλίου η κυρία Λόζινγκ είναι η υπεύθυνη. Θα κάνουμε μια πρώτη ανταλλαγή απόψεων σήμερα. Θα κάνουμε μια πρώτη συζήτηση και στην επόμενη συνεδρίαση της Επιτροπής μας θα έχουμε και το κείμενο και θα κάνουμε την πραγματική συζήτηση. Θα κάνουμε μια αρχική συζήτηση απλώς, εισαγωγική. Κυρία Λόζινγκ. Αγαπητοί συνάδελφοι, στις προηγούμενες συζητήσεις μάθαμε πόσο επίκαιρο είναι το θέμα αυτό και πόσο είναι αναγκαίος ο έλεγχος των εξαγωγών όπλων. Συμφωνούμε όλοι ότι από ηθική αλλά και από πλευρά ασφαλείας και από πλευράς αναπτυξιακής ε, είναι ιδιαίτερα σημαντικό και επίκαιρο το θέμα αυτό. Και πιστεύω ότι και περαιτέρω η εξέταση του θέματος αυτού θα είναι συνενετική. Οι χώρες της Ένωσης συνολικά είναι ο μεγαλύτερος εξαγωγέας όπλων, άρα έχουμε και πολύ μεγάλη υπευθυνότητα να κάνουμε ό,τι μπορούμε για να διασφαλίσουμε ότι τα όπλα που εξάγονται και τα άλλα υλικά πολέμου να μην πέφτουν σε λάθος χέρια. Και αυτό το συζητήσαμε ήδη. Γι' αυτό τον λόγο έχει τεράστια σημασία σε ευρωπαϊκό επίπεδο να υπάρχει ένα λειτουργικό και αποτελεσματικό σύστημα ελέγχου των εξαγωγών όπλων που να εγγυάται τους προαναφερθέντες στόχους. Και εδώ δεν νομίζω ότι υπάρχουν ε, διαφορές απόψεων. Αυτή η συνένεση αντανακλάται και στο ότι το Δεκέμβριο του 2008 υπήρξε αυτή η κοινή θέση για τον έλεγχο της εξαγωγής στρατιωτικής τεχνολογίας και όπλων και στρατιωτικού εξοπλισμού με αυτόν τον τρόπο έγιναν δεσμευτικά νομικά τα 8 κριτήρια που πρέπει να ισχύουν, που μπορεί να είναι βάση καλύτερα για να απαγορευτούν οι εξαγωγές ή να ανασταλούν. Είναι ένα σημαντικό βήμα προς την σωστή κατεύθυνση, γιατί αυτά τα 8 κριτήρια περιλαμβάνουν πολύ βασικά θέματα όπως ο βασμός των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, εάν υπάρχουν συγκρούσεις στην περιοχή όπου εξάγονται, αλλά και κατά πόσον είναι συμβατή η αγορά αυτών των όπλων με την ανάπτυξη της περιοχής στα κριτήρια αυτά, κατά τη γνώμη μου, καλύπτουν πολλά θέματα. Αν και στο ΑΕΒ σημείο οπωσδήποτε θα μπορούσε να υπάρξει κάποια βελτίωση των λεπτομεριών. Για παράδειγμα θα μπορούσαμε να σκεφτούμε το κριτήριο 8 κατά πόσον είναι συμβατά με την ε, ανάπτυξη θα πρέπει να αναβαθμιστεί. Αλλά το κύριο πρόβλημα για μένα είναι αλλού. Ότι ε, έχουμε και συνεχίζουμε να παρατηρούμε ότι συνεχίζονται να γίνονται εξαγωγές όπλων που όσο καλή διάθεση και αν έχει κανείς δεν, μπορούν να θεωρηθεί, δεν μπορεί να θεωρηθεί ότι σέβονται αυτά τα χωροκριτήρια κριτήρια και μάλιστα τα παραβιάζουν. Για παράδειγμα, μεταξύ του 2001 και του 2009 εξά, ε, ε, εξήγε η ε, Ένωση 50 δισεκατομμύρια όπλα προς τις περιοχές που υπάρχουν συγκρούσεις της Μέσης Ανατολής και της Βόρειας Αφρικής. Και στο 2010 50 δισεκατομμύρια δολάρια όπλα. Και επίσης ορισμένες φορές παρατηρήσαμε ότι οι εξαγωγές των γερμανικών όπλων, την οποία εξετάσαμε, διαπιστώσαμε το 2011 δόθηκαν πάνω από 5.800 άδειες εξαγωγής ε, σε 76 χώρες που δεν μπορεί να θεωρηθεί ότι πληρούν αυτά τα κριτήρια. Αυτό είναι 30% των συνολικών εξαγών όπλων της Ομοσπονδιακής Γερμανίας. Είναι προφανές λοιπόν ότι τα 8 αυτά κριτήρια δεν εφαρμόζονται όπως ακριβώς είχε αρχικά προβλεφθεί και όπως όλοι θα επιθυμούσαμε. Πόρισμα. Προφανές κατά τη γνώμη μου. Με βάση αυτό το πλαίσιο χρειάζεται οπωσδήποτε να αναλάβουμε πρωτοβουλίες ούτως ώστε το σύστημα αυτό ελέγχου των εξαγωγών να εφαρμοστεί με πιο αποτελεσματικό τρόπο. Καθήκον λοιπόν του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και της έκθεσή μου είναι να κάνουμε προτάσει προς αυτή την κατεύθυνση. Για αυτό το σκοπό πρέπει πρώτον να αναρωτηθούμε τι επιτρέπει να συνεχίζονται εξαγωγές που αντιτίθενται σε αυτά τα οκτώ κριτήρια. Κατά τη γνώμη μου υπάρχουν δύο λόγοι. Πρώτον, η ερμηνεία και εφαρμογή των 8 κριτηρίων αυτών εξακολουθεί να γίνεται από τα κράτη-μέλη. Αυτό οδηγεί σε πολύ διαφορετικές καταστάσεις για την κατάσταση, για παράδειγμα, των ανθρωπίνων δικαιωμάτων σε μια χώρα και αυτό επηρεάζει τη χορήγηση ή μη της ε, άδειας εξαγωγής. Κατά τη γνώμη μου υπάρχει ανάγκη να δράσουμε ταχύτατα. Πρέπει στόχος μας να είναι μια ομοιογενής ερμηνεία του πνεύματος και του γράμματος αυτών των 8 κριτηρίων. Αν δεν γίνει αυτό, θα συνεχίσουμε να θεωρούμε ότι τα οικονομικά συμφέροντα είναι πολύ πιο σημαντικά από, την, από το σεβασμό αυτών των 8 κριτηρίων. Παρά το ότι στο άρθρο 10 της κοινή θέση εκπεφρασμένα αποκλείεται αυτό το ενδεχόμενο. Όπου λέγεται και παραθέτω, τα κράτη-μέλη μπορούν με ενδεχομένως για κάποιες εξαγωγές να λάβουν υπόψη την οικονομική, βιομηχανική, κοινωνική και πολιτική σημασία των ε, εξαγωγών, αλλά αυτοί οι παράγοντες δεν θα πρέπει να επηρεάζουν και να θίγουν την εφαρμογή των 8 προαναφερθέντων κριτηρίων. Αυτά λέει το άρθρο 10. Ο δεύτερος λόγος για την όχι βέλτιστη εφαρμογή των 8 κριτηρίων, κατά τη γνώμη μου, έχει να κάνει με την ελλειπή αποτίμηση της ε, μέχρι τούδια πρακτικής εξαγωγών. Και εδώ υπάρχουν κάποιες δυνατότητες εξαγωγής για την ετήσια έκθεση που γίνεται για τις εξαγωγές των μονομένων κρατών μελών. Θα έπρεπε λοιπόν να δημοσιεύονται εγκαίρως αυτές οι εκθέσεις και να υπάρχει και μια συνόψη των κυρίων πορισμάτων όπου να φαίνονται οι αλλαγές και οι τάσεις ε, σε σχέση με το προηγούμενο έτος. Αυτή η έκθεση λοιπόν, εάν διαμορφωνόταν έτσι, θα ήταν πολύ πιο χρήσιμη. Επίσης, σημαντικό είναι να υπάρχει και ένα νέο σύστημα εκπόνησης αυτών των εκθέσεων που να αναφέρει ποια στοιχεία, με ποια μορφή πρέπει να δίδονται από όλα τα κράτη και να δίδονται πλήρως. Γιατί μέχρι στιγμής δεν ε, χορηγούν όλα τα κράτη πλήρη στοιχεία. Το 2010 με βάση το Ινστιτούτο για την έρευνα ε, για την ειρήνη στην Ευρώπη, μόνο 23% των δεδομένων είχαν υποβληθεί. Χρειάζεται λοιπόν μεγάλη βελτίωση. Γιατί λοιπόν μέχρι στιγμής παραβιάζονται τα 8 κριτήρια. Γιατί δεν αποτιμάται σωστά η πολιτική και πρακτική των κρατών. Γι' αυτό οι εκθέσεις θα έπρεπε στο μέλλον να συμπεριλαμβάνουν μια τέτοια αποτίμηση της πρακτικής των κρατών που να μας δίνει στοιχεία εάν και σε τι βαθμό η πρακτική των μεμονωμένων κρατών της Ένωσης τηρεί το πνεύμα και το γράμμα των 8 κριτηρίων. Από την άλλη μεριά όμως ε, οι επιχειρήσεις θέλουν να διευκολύνουν και κάνουν, ε, υποβάλλουν αιτήματα όπου λένε ότι, ότι επειδή μειώνεται η εσωτερική ζήτηση πρέπει να το, το αντιμετωπίσουν αυτή τη μειωμένη εσωτερική ζήτηση με αύξηση των εξαγωγών. Αυτό μπορεί να σημαίνει αύξηση των εξαγωγών σε περιοχές που υπάρχουν συγκρούσεις όπως η Μέση Ανατολή, η Βόρεια Αφρική. Αλλά εδώ έχουμε ήδη δει τι μοιραίε επιπτώσει μπορεί να έχει η εξαγωγή όπλων σε αυτέ τι περιοχέ. Γι' αυτό χρειάζεται πιο αποτελεσματικό σύστημα ελέγχου των εξαγωγών όπλων, όπω προτείνω, θα προτείνω στην έκθεσή μου. Και ελπίζω, συνάδελφοι, να με υποστηρίξετε στι προσπάθειέ μου. Ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστούμε για την παρουσίαση που ήταν πλήρης, πυκνή. Ο Κρίστοφ Λίσεκ είναι ε, σκιώδης του ΕΛΚ. Θα μας μιλήσει τώρα. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Η κυρία Λέζινγκ παρουσίασε με ενδιαφέροντα τρόπο το θέμα. Την ευχαριστώ. Είναι κρίμα που δεν έχουμε ένα έγγραφο εργασίας να βασιστούμε σε αυτό. για τη σημερινή συζήτηση. Αλλά ετοιμάζεται από την κυρία Λέζινγκ, από ό,τι κατάλαβα, αυτό το κείμενο και το περιμένουμε. Περιμένουμε και προσβλέπουμε στη συνεργασία. Περιμένουμε να συζητήσουμε πιο ενδελεχώς το θέμα μαζί σας, κυρία Λέζινγκ. Κυρία Λέζινγκ, μας είπατε ποια είναι τα θέματα, ποιες είναι οι προκλήσεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αξίζει να πούμε ότι τυπικά η Ευρωπαϊκή Ένωση ως οργανισμός δεν εξάγει όπλα. Εξάγουν τα κράτη-μέλη. Και σε ορισμένε περιπτώσεις δεν εξάγουν καν τα κράτη-μέλη. Διότι η βιομηχανία όπλων ε, ανήκει στον ιδιωτικό τομέα σε πολλά Δεν εξάγει δηλαδή το κράτος επίσημα όπλα. Εξάγουν κάποιες εταιρείε. Φυσικά, αυτές οι ιδιωτικές εταιρείε ε, ορμώνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Έχουν έδρα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Μην ξεχνάμε ότι οι εξαγωγές όπλων ήταν πάντα ένα αμφι... αμφίσιμο θέμα, ένα επίμαχο θέμα και συμφωνώ βεβαίω ότι κάποιοι κανόνε θα πρέπει να γίνουν πιο αυστηροί και κάποιοι κανόνε θα πρέπει να γίνονται σεβαστοί κατά την εξαγωγή όπλων. Αλλά όμω μην ξεχνάμε ότι στα κράτη-μέλη τα, τα όπλα δεν είναι μόνο αντικείμενο εμπορίου. Ε, η βιομηχανία αυτή δημιουργού θέσεις απασχόλησης. Ε, Δεκάδες χιλιάδες άτομα δουλεύουν σε αυτόν τον κλάδο. Στην ε, Πολωνία, βέβαια εμείς δεν εξάγουμε πολλά όπλα, δεν εξάγουμε από την Πολωνία, κι όμως πολλοί Πολωνοί, δεκάδες χιλιάδες ε, Πολωνοί εργάζονται στον κλάδο αυτό. Μην το ξεχνάμε αυτό. Από την άλλη υπάρχει τεράστιος ανταγωνισμός μεταξύ των ε, διαφόρων χωρών. Αν προσθέσετε και τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι εξαγωγές όπλων συνολικά είναι μια πολύ επικεντής επιχείρηση. Ε, η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι ένας μεγάλος ανταγωνιστής των ΗΠΑ στον τομέα αυτό. Το μερίδιό μας στις εξαγωγές όπλων είναι μεγαλύτερο από της Ρωσίας. Αν δεν εξάγαμε όπλα, ας πούμε σε κάποιες περιπτώσεις, ποιος θα σε αυτήν την περίπτωση, αμερικανικές και ρωσικές εταιρείες στη θέση μας. Και θα κάλυπταν πάρα αυτό το κενό που θα αφήναμε εμείς. Περιμένουμε και το κείμενο πάντως, γιατί είναι χρήσιμο. Το θέλουμε το συντομότερο δυνατόν και είμαι έτοιμος να συνεργαστώ με την κυρία Λέζιν για το θέμα αυτό. Ευχαριστώ. Ο επόμενο ομιλητή. Ευχαριστώ. Θα ήθελα και εγώ να ευχαριστήσω την εισηγήτρια για τα κέρια λόγια της. Υπάρχουν κάποια ερωτήματα παρόλα αυτά. Η αρχή που επικαλέστηκε οι αρχές που επικαλέστηκε είναι απόλυτα βάσιμες και εφαρμόζονται σε περίπτωση σύγκρουση, σύγκρουσης πολλών, μεταξύ πολλών κρατών. Δηλαδή για τις διεθνές σειράξεις πολύ σωστές είναι αυτές οι αρχές. Το θέμα είναι τι κάνουμε απέναντι στις νέες μορφές συγκρούσεων. Γιατί οι σημερινέ σειράξει, οι σημερινοί πόλεμοι είναι τελείω διαφορετικοί από του πολέμου τη δεκαετίας του 70 ή του 80. Έχουμε ενδοκρατικές συγκρούσεις σήμερα. Ε, εάν χρησιμοποιήσουμε αυτές τις αρχές, αφήνουμε ε, ανυπεράσπιστες ε, κάποιες κοινότητες. Νταρφούρ, Μαλή, Ανατολικό Κονγκό, υπάρχουν κοινότητες που θα τις αφήναμε στην τύχη τους. Στη Συρία, ας πούμε. Δηλαδή, αυτές οι αρχές και αυτή η συνθήκη καλύπτει όλες τις περιπτώσεις όπου διάφορα, διάφορες εθνότητες, διάφορες κοινότητες εσωτερικών ως κράτους ε, είναι σε πόλεμο. Ε, έχετε δίκιο σε αυτά που είπατε. δεν εμπνευστήκαμε αρκετά από το έγγραφο ευθύνη για την προστασία. Responsibility to protect. Σε αυτό το σχέδιο συνθήκης υπάρχει ένα κενό. Μήπως θα πρέπει να πάμε πιο μακριά. Μπορούμε να απαντήσουμε σε αυτά τα ερωτηματικά. Όπου πολύ συχνά το διεθνές δίκαιο αφήνει ανθρώπους να πεθαίνουν χωρίς να τους υπερασπίζεται κανείς. Εδώ δεν υπάρχουν απαντήσεις. Αισθάνομαι ότι κάτι λείπει. Ο επόμενος ομιλητής. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Νομίζω ότι πρέπει να μιλάμε για συνεργασία ε, σε ό,τι αφορά τον έλεγχο των εξαγωγών όπλων. Παναλαμβάνω γιατί υπήρχε πρόβλημα με τη γερμανική διερμηνία. Πρέπει να συζητάμε τη συνεργασία ε, στο τομέα των εξαγωγών όπλων. Γιατί πρέπει να έχουμε κάποιου κοινού κανόνες. Το εμπόριο όπλων από μόνο του δεν είναι κάτι το κακό, εφόσον υπάρχει κάποιο έλεγχος. Είναι σημαντικό αυτό το εμπόριο για την ασφάλεια της Ευρώπης και για την ασφάλεια της χώρας μου, της Φιλανδίας. Υπάρχει το νόμιμο εμπόριο όπλων και εκεί δεν πρέπει να βάζουμε προσκόμματα αλλά πιστεύω ότι πρέπει να υπάρχουν αυστηρότεροι έλεγχοι στο παράνομο εμπόριο. Σε αυτή την πρώτη συζήτηση που κάνουμε σήμερα, θέλω να πω ότι προσβλέπω σε μια συνεργασία με την κυρία Λέζη, Ελπίζω να μπούμε και σε λεπτομέρειες, να συζητήσουμε τις λεπτομέρειες του κειμένου εν ευθέτω χρόνο. Το θέμα είναι πολύ ευρύ είναι πολύ περίπλοκο. Και δεν νομίζω ότι θα είναι εύκολο να συμφωνήσουμε στην υποεπιτροπή μας ε, τόσο εύκολα. Θα πρέπει να συζητήσουμε πολύ. Ευχαριστώ. Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης. Ο κύριος Ντελαπιάτσα. Ε, θα μιλήσω αγγλικά. Είμαι πρόεδρος της ομάδας εργασίας του Συμβουλίου που ασχολείται με την εξαγωγή συμβατικών όπλων, COARM, που είναι υπεύθυνη δηλαδή και για την, το συντονισμό και την εφαρμογή της κοινή θέση μεταξύ των κρατών μελών και να προετοιμάσει την ετήσια έκθεση που αναφέρθηκε από την κυρία Λέζινγκ. Θα ήθελα να προσθέσω δύο στοιχεία στη συζήτηση, ελπίζω να σας βοηθήσουν ε, για να προετοιμάσετε και την έκθεση που η Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης περιμένει, γιατί θέλουμε να συνεργαστούμε και μπορούμε να σας δώσουμε και πληροφορίες, ούτω ώστε το Κοινοβούλιο να είναι σε θέση να παίξει το ρόλο του και να αναλάβει τις ευθύνες του. Η κοινή θέση υιοθετήθηκε το 2008 ως ε, εργαλείο μέσω της ΚΠΑ, αποτέλεσε σημαντική βελτίωση στον τρόπο με τον οποίο συντονίζουν και εναρμονίζουν τα κράτη-μέλη τις πολιτικές ελέγχου του εμπορίου όπλων. Η κοινή θέση βέβαια από μόνη της δεν μπορεί να κάνει κάτι που δεν θέλαμε να κάνει. Υπάρχουν 8 κριτήρια, ευραία, καλύπτουν διάφορα θέματα. Από νομικής άποψης είναι πολύ ευραία τα κριτήρια και η κοινή θέση προσδιορίζει σαφώς ότι, ότι η εφαρμογή και η ερμηνεία των κριτηρίων είναι θέμα κρατών μελών. Είναι βασικό στοιχείο. Εγώ δεν θεωρώ την ελάττωμα. Μην το ξεχνάμε αυτό. Όταν αξιολογούμε τι κάνουν τα κράτη-μέλη εφαρμόζοντας την κοινή θέση, μην ξεχνάμε αυτό το στοιχείο. Οι εξαγωγικές πολιτικές των κρατών μελών, το αν είναι επαρκώς υπεύθυνε. αυτό είναι ένα θέμα, βεβαίως πολύ σημαντικό, αλλά δεν συνδέεται στενά με την ε, εφαρμογή της κοινή θέση κατά ανάγκη. Ε, το θέμα αυτό είναι όχι πολιτική απόφαση, το θέμα της κοινή θέση δηλαδή, ε, είναι θέμα ύπαρξης κάποιων διαδικασιών. Κάτι άλλο που είναι σημαντικό, θέλω να υπενθυμίσω. Αν τα κράτη-μέλη δεν πρέπει να εξάγουν κανένα όπλο ή οπλισμό σε καμία τρίτη χώρα που παραβιάζει τα ανθρώπινα δικαιώματα, τότε δεν θα υπήρχε καμία εξαγωγή. από πολλά κράτη-μέλη. Ίσως τελικά μακροπρόθεσμα αυτό πρέπει να πετύχουμε. Αλλά αυτό που λέει στην πραγματικότητα η κοινή θέση είναι ότι κάθε εξαγωγή θα πρέπει να αξιολογηθεί κατά περίπτωση. Μπορεί να σας μοιάζει τεχνικό αυτό. Αυτό τι σημαίνει. Όταν μια εθνική αρχή πρέπει να αποφασίσει αν θα δώσει άδεια σε μια εξαγωγή, θα πρέπει να λάβει ε, υπόψη κάποια στοιχεία, το είδο των όπλων που μπορούν να εξαχθούν, τον όγκο τους, το είδος της χρήσης, το χρήστη, με βάση τις δηλώσεις των ενδιαφερομένων. Και αν τις δηλώσεις αυτές μπορούμε να τις ε, εμπιστευτούμε. Αυτή την πολιτική αξιολόγηση πρέπει να την κάνει η Εθνική Αρχή. Αυτό τι σημαίνει, ότι να πουλάμε ας πούμε τάγκ σε μια χώρα του κόλπου δεν είναι το ίδιο με το να πουλάμε μικρά ας πούμε όπλα και ελαφριοπλισμό σε χώρες του κόλπου. Αυτό πρέπει να το λάβουμε υπόψη μας. Επίσης, υπάρχουν και κυρώσει στην Ευρωπαϊκή Ένωση που μπορούν να εφαρμοστούν όταν είναι αυτό σκόπιμο πολιτικά. Η ετήσια έκθεση, τελευταίο σημείο. Δεν ξέρουμε αν θα είμαστε εμπρόθεσμοι, αλλά θα πρέπει να έχουμε όλα τα στοιχεία και από τα 27 κράτη-μέλη και μόνο τότε θα είμαστε έτοιμοι να την ετοιμάσουμε. Θα προσπαθήσουμε μέσα στην επόμενη χρονιά να είμαστε έτοιμοι δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή ε, κάποια χώρα που δεν συμμορφώθηκε με τις υποχρεώσεις ε, σύνταξης έκθεσης. Αυτό που είπε η κυρία Λέζιν αφορούσε τις πραγματικές εξαγωγές που γίνονται και όχι μόνο τις άδειες εξαγωγών. Και τα δύο, και οι δύο κατηγορίες θα πρέπει να αναφέρονται. Εγώ θα σταματήσω, είμαι στη διάθεσή σας και εγώ και οι υπηρεσίες μου να συνεργαστούμε με την υποεπιτροπή σας για το θέμα αυτό. Merci. Ευχαριστώ. Ο κύριος Γκέρινγκς και εν συνεχεία η κυρία Λόιζινγκ για τα τελικά της σχόλια. Ας είμαι πιο ακριβής. Ο εξοπλισμός των δυνάμεων που είναι αντίθετες στο συριακό καθεστώς. Συνάδει, είναι αντίθετος με τις οχτώ αρχές που ακούσαμε. Δηλαδή, ο σεβασμός αυτών των οχτώ κριτηρίων ε, γίνεται ε, για όλο τον οπλισμό των ομάδων που πολεμούν για την ελευθερία τους. Μπορούν δηλαδή να προστατευθούν με την εφαρμογή αυτών των οχθοκριτηρίων κριτηρίων, αγοράζοντας τα όπλα που χρειάζονται. Λαμβάνει υπόψη αυτή η ε, συνθήκη την κατάσταση, τη φύση των ε, συγκρούσεων που λαμβάνουν χώρα σήμερα, που είναι εντός ενός κράτους. Νομίζω ότι αυτά τα κριτήρια ισχύουν όταν οι πόλεμοι γίνονται μεταξύ κρατών. Αλλά δεν λαμβάνουν υπόψη τι συμβαίνει όταν το πρόβλημα είναι στο εσωτερικό ενό κράτου. Και ζητώ συγγνώμη, αλλά η σύγχυση βασιλεύει στο εσωτερικό ενός κράτους μεταξύ διαφόρων κοινοτήτων ή εθνοτήτων κτλ. Για τη Συρία. Η πολιτική της Ένωσης προβλέπει ε, κυρώσεις και εμπάργκο ε, για την εξαγωγή όπλων στη Συρία. Η κοινή θέση δεν έχει καμία σχέση Υπάρχουν άλλα μέτρα που προβλέπονται. Υπάρχουν κυρώσει που, που επιβάλλουν εμπάργκο στην πώληση όπλων στη Συρία. Τώρα, θεωρητικά, εάν δεν υπήρχε εμπάργκο, πώς θα εφαρμοζόταν η κοινή θέση. Στην κοινή θέση υπάρχουν πολλά στοιχεία. Όχι μόνο ο κίνδυνος ε, συγκρούσεων μεταξύ κρατών, αλλά και η περιφερειακή σταθερότητα πρέπει να τα λάβουμε υπόψη μας ε, ανάλυοντας μια κατάσταση. Αλλά η εφαρμογή αυτών των ε, αρχών είναι ευθύνη των κρατών μελών και η ερμηνεία αυτών των αρχών. Με βάση την εμπειρία μας προκύπτει ότι μερικές φορές τα κράτη-μέλη φτάνουν σε συμπεράσματα τα συμπεράσματα στα οποία φτάνουν τα κράτη-μέλη είναι τελείως διαφορετικά από κράτος σε κράτος. Δεν μπορώ να σας δώσω σαφείς απαντήσεις σε αυτά τα ερωτήματα, κυρία Λέζη, για τα τελευταία τη σχόλια. Νομίζω ότι έχουμε μπει σε μια πολιτική συζήτηση. Δεν θα ήθελα να περάσω σε όλες τις λεπτομέρειες, αλλά μια απάντηση. Όπλα σε, εποχές, σε περιοχές όπου υπάρχει κρίση απαγορεύεται. Στην έκθεσή μου ασχολούμαι με την εφαρμογή των κριτηρίων της κοινή άποψης δεν θα συζητήσω τώρα το α ή το β κριτήριο. Δεν είναι αντικείμενο της εκθεσής μου αυτό. Και μία απάντηση ακόμη. Εξαγωγές όπλων σε περιοχές κρίσεων προς δυνάμεις των Ηνωμένων Εθνών που είναι εκεί για να προστατεύσουν κάποιους, δεν απαγορεύεται φυσικά. Για αυτά που είπε ο κύριος Λίζεκ. Φυσικά πολλά θέματα που θα περιληφθούν στην έκθεσή μου σχετίζονται συμφέροντα των κρατών μελών σε σχέση με τις προϋποθέσεις των ε, οκτώ κριτηρίων. Πρέπει δηλαδή να τα συνεκτιμήσουμε αυτά. Μας ενδιαφέρει να δούμε αν εφαρμόζονται τα κριτήρια. Είπατε, μα δεν ε, εξάγουν κράτη εξάγουν ε, επιχειρήσεις. Αλλά οι επιχειρήσεις για να εξαγάγουν χρειάζονται κρατικές άδειες. Αυτό είναι το θέμα της εκθεσής μου. Από αυτά που είπε, για αυτά που είπε η Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης, βεβαίως πρέπει να τα συζητήσουμε πιο αναλυτικά από κοινού δεν είναι δυνατό να γίνει τώρα στα πλαίσια της συνεδρίασης. Θα ήθελα να περιοριστώ σε αυτές τις απαντήσεις ε, σε αυτή τη φάση, διότι η συζήτηση τώρα για την έννοια που έχουν τα επιμέρους κριτήρια δεν είναι αντικείμενο της έκθεσής μου. Ευχαριστώ για αυτήν την πρώτη ανταλλαγή απόψεων θα επανέλθουμε όταν θα έχουμε το πρώτο σχέδιο έκθεση στην επόμενη συνεδρίασή μας. Αν δεν υπάρχουν άλλα θέματα, κλείνει η συνεδρίαση και η επόμενη συνεδρίασή μας θα είναι στις 20 Φεβρουαρίου, αλλά θα έχουμε την ακρόαση του Γάλλου Υπουργού Εξωτερικών που δεν είναι Δευτέρα στην ΑΦΕΤ θα γίνει στο Στρασβούργο κατά την Ολομέλεια αρχές Φεβρουαρίου. Είμαστε σε συνεννόηση